Uh, uh, ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω. Μία συνεδρίαση θα έχουμε της Επιτροπής μας αυτή την εβδομάδα. Να σας πω κάτι πρακτικό πριν να ξεκινήσουμε. Όσοι θέλουν να ακούσουν ε, τη γερμανική μετάφραση, μας είπαν οι ότι το κανάλι 1 ε, δεν ε, λειτουργεί σήμερα, έχει αποσυνδεθεί. Έτσι λοιπόν για τη γερμανική μετάφραση θα πρέπει να ακούτε το κανάλι 27. Έτσι λοιπόν θα δώσω το λόγο στους γερμανούς συναδέλφους για να κάνουμε μια δοκιμή. Και αν δεν δουλεύει το κανάλι 27, τότε να μου κάνετε ένα νόημα και θα προσπαθήσω να επιλύσω την κατάσταση στη συνέχεια. Κανάλι 27 λοιπόν για τα γερμανικά, για σήμερα το απόγευμα. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα ημερική διάταξη και θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στη μήνυ ακρόαση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και θα προεδρεύσει η Αντιπρόεδρος η κυρία Μπερνατέ Βερνιό μαζί με την ε, κυρία Κόμη. Προεδρεύσουμε λοιπόν για το θέμα αυτό και θα αναφερθώ στη συνέχεια. Πριν να προχωρήσουμε στα δύο προηγούμενα θέματα, ε, στα δικαιώματα και στην προστασία των καταναλωτών. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους για το εξή Το Προεδρείο της Επιτροπής είχε ένα πολύ χρήσιμο γεύμα με τον καθηγητή Μάριο Μόντι. Νομίζω όλοι θα έχετε δει την ανακοίνωση ότι ο καθηγητής Μόντι ε, ανατέθηκε στον κύριο Μόντι από τον ε, πρόεδρο της Κομισιόν Μπαρόσου μια ειδική αποστολή να επικεντρωθεί ε, στο μέλλον της ε, νέας αγοράς. Και καθώς εμείς είμαστε η Ειδική Επιτροπή, η κυρία Επιτροπή, με το θέμα αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγώ ανέλαβα την πρωτοβουλία να σας προτείνω να γράψουμε μια επιστολή στον κύριο Μόντι. Ε, τώρα έχει συναντήσει ένα, ένα αριθμό μελών και αυτή λέει μελέτη είναι προσωπική αποστολή Εμεί αναμένουμε να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του χρόνου. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα στρατηγικό έγγραφο και νομίζω ουσιαστικά προσπαθεί ο πρόεδρος Κομισιών Κομισιόν να πλαισιώσει την εργασία των μελών της Κομισιόν και έτσι νομίζω ότι είναι θεμελιώδες και η εργασία εδώ στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, ελπίζω ότι όλοι υποστηρίζετε ότι εγώ και το Προεδρείο ήρθαμε πολύ γρήγορα σε επαφή με τον κύριο Μόντι, γιατί αν πρέπει, πρέπει να είμαστε από την αρχή ε, στη διαδικασία για να επηρεάσουμε. Και μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτό ε, και θέλει να ακούει τις ιδέες μας. Και θα διανύμουμε, μάλλον συγγνώμη, έχουμε διανύμει την επιστολή, ένα αντίγραφο της επιστολής, ε, από τον κύριο προς τον κύριο Μόντι, όπου αναφέρεται ξεκαθαρά η εντολή που του δίνεται. Όμως νομίζω ότι το πεδίο το, της εργασίας του κ. Μόντι θα εστιάσει στο να υπάρχουν ωφέλη από την ενιαγορά αγορά για όλους τους Ευρωπαϊκούς πολίτες και πώς θα βελτιώσουμε ε, αυτά τα ωφέλη. Και επίσης νομίζω και το θέμα της οικονομίας θα είναι σημαντικό στη συζήτηση ο κύριος ε, Μόντι προσφέρθηκε να μας συναντήσει στο Στρασβούργο του Δεκεμβρίου, αν συμφωνήσουν και οι συντονιστές. Και φυσικά, αν τελικά συμφωνήσουμε, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Γιατί θα... μπορούμε uh, λοιπόν, να προχωρήσουμε. Uh, can I ask formally for να ζητήσω, αν συμφωνείτε, με την έγκριση της της διάταξης. Um, Uh, Επίσης, έχουμε μοιράσει τα πρακτικά για τις 4 και 5 Νοεμβρίου 2009. Μπορώ να ζητήσω την έγκριση των πρακτικών. Ευχαριστώ. Right. Let's now move on to, uh... Να προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω συζήτηση για αυτό το σημαντικό project για τα δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι η κύρια νομοθετική πρόταση που έχουμε επιτάπτει σε αυτή τη στιγμή. Και θα δώσω το λόγο σε λίγο στον Άντριο ε, Σφαμπ και έχουμε και τους και τη εδώ, κυρία Κάπ, κύριε Ρόσφορ, κύριε Τούρνερ, νομίζω ο κ. Μιλάνε δεν είναι εδώ. Έχουμε επίσης εδώ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, την Τζοζέπη Μόντι. Όχι, συγγνώμη. Κάποιος άλλος συνάδελφος θα μιλήσει εκ μέρου της Κομισιόν. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν αφού θα έχουμε ανταλλαγή απόψε. Και έχουμε επίσης και τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας τη Σουηδικής Προεδρίας. Κύριε Στάλιν, αν θέλετε να συνεισφέρετε στο μέλλον, είστε πρόσδεκτος. Όλοι λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι είναι εδώ. Είχαμε μία δημόσια κρόταση στις 29 Σεπτεμβρίου και είχαμε και έναν επίσημο έγγραφο από την Κομισιόν που ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι ο κύριος Σβάπ θα μιλήσει για το χρονοδιάγραμμα και πότε σκοπεύουμε να έχουμε μία ανακρόση και θα μας πει πώς προχωρούν οι εργασίες. Παρακαλώ, Ανδρέας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που σήμερα μπορούμε να ε, συζητήσουμε την οδηγία αυτή με κάπως πιο διαρθρωμένο τρόπο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης που ε, έχουν συνεργαστεί επικοδομητικά για πολύ δύσκολα ζητήματα. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στα άρθρα 1 έως 3 και στις επόμενες συζητήσεις θα συζητήσουμε τα 4 και 5. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κέπχαρτ, τον κύριο Τούνες, για τις πολύ καλές προτάσεις τους για τροπολογίες. Θα παρουσιάσουν ήδη τις τροπολογίες τους, αλλά στόχος μας είναι μαζί να λύσουμε, να εξετάσουμε όλα τα δύσκολα θέματα της οδηγίας αυτής και να τα συγκεντρώσουμε σε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο θα έχουμε ολοκληρώσει όταν θα έχουμε ε, συζητήσει ε, εις βάθος όλα τα ζητήματα. Και στο έγγραφο εργασία αυτό θα εξετάσουμε ξεχωριστά το κάθε κεφάλαιο. Δεύτερον, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή Δικαιοσύνη επίση ε, είχε μια. Η Νομική Επιτροπή είχε μια συζήτηση για το ε, θέμα αυτό. Έχουν αναθέσει μια, την διεξαγωγή μια μελέτη για το ζήτημα αυτό. Και η συζήτηση που έγινε για τη μελέτη αυτή είχε ως αποτέλεσμα κυρίως μια επίκριση ότι το σχετικό πλαίσιο δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς στην πρόταση της Επιτροπής. Ε, φυσικά εμείς θα φροντίσουμε ε, στο βαθμό που είναι δυνατόν να ενσωματωθεί διότι φυσικά όλοι ενδιαφέρονται τα κράτη-μέλη μακροπρόθεσμα πρόθεσμα να ενδιαφερθούν για αυτό το, το, το εγχείρημα εναρμόνισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό σημαντική πίεση χρόνου έχει εκπονήσει μια επισκόπηση του κεφαλαίου 1 και εξετάζει την ε, παρούσα κατάσταση της ελάχιστης ε, εναρμόνισης ε, σε σχέση με την μελλοντική κατάσταση της μέγιστης εναρμόνισης. Και θα ήθελα τώρα, πολύ σύντομα, να σας αναφέρω κάποια σημαντικά δύσκολα ζητήματα στα κεφάλαια 1 έως 3. Στο κεφάλαιο 1 θα ήθελα Μάλλον θέλω πρώτα να αναφερθώ στο, ε, ναι, ε θέλω να αναφερθώ στο, ε, στο άρθρο 2, σημείο 5. Ε, δεν θέλουμε να έχουμε στο πεδίο σε μόνο τα αγαθά, αλλά και τις υπηρεσίες στην οδηγία αυτή για την προστασία του καταναλωτή. Μέχρι στιγμής, η πολυπλοκότητα της της ε, ε, συμπερίληψης των ε, υπηρεσιών έχουν οδηγήσει σε δυσκολίες ότι το 95% των υπηρεσιών στην Ευρώπη παρέχονται σε τοπικό επίπεδο. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και κάποιες, κάποια άλλα σημεία της πρότασης οδηγίας όσον αφορά το θέμα αυτό. Στο 2.12, στο άρθρο 2 σημείο 12. Έχουμε νομοθετική σαφήνεια, αλλά δεν είμαι βέβαιος εάν ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια γενική εικόνα της ε, σημερινής κατάστασης. Υπάρχει το θέμα της εξαίρεσης ε, των δημοσίων προμηθειών, των ε, δημοπρασιών, ε, συγγνώμη, αναφερόμαστε και στο eBay. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτές τις δημοπρασίες δημόσιες. Θα πρέπει οι καταναλωτές ε, να έχουν και σε αυτές τις ε, περιπτώσεις υψηλό επίπεδο προστασίας. Όσον αφορά την συζήτηση για το άρθρο 4 που αποτελεί κεντρικό σημείο της πρώτης οδηγίας αυτής, ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχετε λίγη υπομονή. Το θέμα είναι πώ ε, μπορούμε να διαμορφώσουμε αποτελεσματικά το σύστημα προστασία του καταναλωτή εντό τη Ευρώπη. ώστε και στα 27 κράτη-μέλη τη Ευρώπη να προστατεύονται οι καταναλωτέ. και υπάρχει βέβαια το θέμα τη ελάχιστη εναρμόνιση, τη περίστευσης εναρμόνιση, τη τομιακή εναρμόνιση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εξετάσουμε κάθε υποπαράγραφο της πρότασης οδηγίας ε, για να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους καταναλωτές ε, της Ευρώπης. χωρίς να περιορίσουμε την ευρεία επιλογή αγαθών που έχουν αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές. Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πω ότι η υποχρέωση ενημέρωσης ε, του καταναλωτή που πιστεύω ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί σε όλη την Ευρώπη βελτιώνει τη διαφάνεια και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Ε, γι' αυτό θα επικροτούσαμε κάτι τέτοιο. Αλλά και εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην δυσκολέψουμε τους καταναλωτές. Να λαμβάνουν δηλαδή την ε, τον σωστό όγκο πληροφοριών. Στο παρελθόν, ε, ιδιαίτερα για τις καταναλωτικές πιστώσεις, ε, έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. Μερικές φορές οι καταναλωτές ε, λαμβάνουν υπερβολικά πολλές πληροφορίες που ουσιαστικά τους μπερδεύουν περισσότερο παρά τους βοηθάνε. Όσον αφορά το κεφάλαιο 3... Η συμπερίληψη των ε, αγορών εξ και των ε, αγορών ε, στην πόρτα του καταναλωτή πιστεύω ότι είναι κάτι θετικό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε εξαιρέσεις και για παράδειγμα για τα ευπαθή προϊόντα που εξαιρούνται από την πρόταση οδηγίας της Κομισιόν. Έχω επανειλημμένα πει ότι ε, κάποια ε, γερμανική εφημερίδα θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να την επιστρέψω μετά την αγορά. Μια πολύ γνωστή ε, εφημερίδα της Γερμανίας που δεν είναι πάρα πολύ σοβαρή. Σίγουρα θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα του τύπου και της πώληση στο δρόμο. Όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας, ο τύπος θα πρέπει να επιδείξει υψηλότερα πρότυπα ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει όταν αγοράζει μια εφημερίδα ε, ότι έχει ακολουθηθεί ο κώδικας διοντολογίας. Μήπως όμως θα πρέπει να ε, έχουμε και εδώ παρέκκληση στην οδηγία όσον αφορά το άρθρο 10. Πολλά κράτη-μέλη, πολλές επιχειρήσεις, ε, πολλοί καταναλωτές θα επωφεληθούν εάν απλοποιήσουμε το άρθρο αυτό με τρόπο όμως ώστε το δικαίωμα, η άσκηση του δικαιώματος επαναχώρησης ε, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο να μην ε, καταργηθεί, να μην ε, δυσκολευτεί. Και στο κεφάλαιο 3, στο άρθρο 27, προτείνεται ο καταναλωτής να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δύο εβδομάδων εάν έχει λάβει ένα προϊόν το οποίο δεν του αρέσει και υπολογίζονται και άλλες ε, δύο εβδομάδες από την αποστολή του προϊόντος ε, μέχρι να το λάβει η επιχείρηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο εξής ερώτημα. Εάν με νομικές διατάξεις μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα που, που, τα προβλήματα που ε, ε, συναντάει ο καταναλωτής και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ε, εσωτερική αγορά. διότι το θέμα της επιστροφής των προϊόντων, του δικαιώματος παναχώρησης, δεν είναι μόνο οι προθεσμίες. Έχουμε 27 διαφορετικούς ταχυδρομικούς οργανισμούς στα κράτη-μέλη Εάν λοιπόν ε, το ταχυδρομείο δεν ε, ενεργεί γρήγορα, τότε δεν, είναι, δεν φταίει ο καταναλωτής γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν πιστεύω να το λάβουμε αυτό υπόψη κατά την εξέταση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Και κλείνοντας ε, να πω ότι τις επόμενες όταν συζητήσουμε τις λεπτομέρειες τη οδηγίας αυτές θα πρέπει να εξετάσουμε σε ποια σημεία μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τον καταναλωτή με νομοθετικά μέτρα και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να βοηθήσουμε με άλλους τρόπους για παράδειγμα με την καλύτερη εφαρμογή του νόμου με την καλύτερη, με την καλύτερη επιβολή του νόμου. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα Ευρωπαϊκά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη υπάρχουν αστικοί κώδικες που έχουν διαμορφωθεί ε, σε βάθος χρόνου, θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι σήμερα μπορούμε να εργαστούμε πολύ πιο γρήγορα κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει ε, να μπορούμε να εξηγήσουμε στον καταναλωτή και στις επιχειρήσεις ε, το νέο σύστημα και θα πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα πριν ε, τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία. Αναφέρθηκα στις ε, υπηρεσίες που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει όμω να σκεφτούμε μήπω μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της οδηγίας ε, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογή. Και επίση ε, στο κεφάλαιο 1, Μήπω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όρους από άλλες οδηγίες, Θα πρέπει να πείσουμε τον καταναλωτή ότι είναι μια χρήσιμη οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο και γι' αυτό πιστεύω ότι την επόμενη συζήτηση θα πρέπει να την διεξάγουμε ε, μαζί με τους συναδέλφους από ε, τα κοινοβούλια των ε, Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών. Έχουμε οργανώσει μία συζήτηση με τους συναδέλφους από το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Πρέπει άλλωστε να καταστήσουμε σαφές ότι πολύ λίγες ε, οδηγίες φεύγουν ε, από το Κοινοβούλιο ή υπό τη μορφή που ε, έρχονται στο Κοινοβούλιο. Πάντως θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στις εργασίες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σβάπ για τις πολύ σαφείς εξηγήσεις σας. Ως πρόεδρος να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα τεχνικά ζητήματα για τις 2 Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να έχουμε βίντεο διάσκεψη, επιγραμμική ανταλλαγή απόψεων με τους Γάλλους συναδέλφους και όπως είπατε και το Βρετανικό Κοινοβούλιο θέλει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών του στις 23 Φεβρουαρίου. Έχουμε οργανώσει αυτήν την ε, δεύτερη ακρόαση. Να δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις συζητητές. Είναι ανοιχτό ο καταλόγος των ομιλητών για όποιον άλλον θέλει να παρέμβει. Η κυρία Κέπχαρτ, ο κυριο Ρόσφορτ, η κυρία Τούρνερ και ο κύριος Τριανταφυλλίδη. Εάν θέλει άλλος να ε, μιλήσει, να το πει η κυρία Κέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σφάμπ για την παρουσίαση. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά θέματα, παρόλο που πολλά τα έχουμε ήδη συζητήσει και επεξεργαστεί. Ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί επιμηκύνθηκε λίγο η περίοδος επεξεργασίας. Υπάρχουν πολλά λοιπόν που πρέπει ακόμα να εντοπίσουμε, που υπάρχουν ακόμα δυσκολίες, που υπάρχουν πλέον εκτήματα και τι απαντήσεις ε, μπορούμε να δώσουμε σε αυτό τον τομέα. Βεβαίως και το θέμα είναι περίπλοκο και διαβάζοντας την πρόταση είδα ότι υπάρχουν προβλήματα και όσον αφορά τα παιδιά εφαρμογής και όσον αφορά τους ορισμούς. Καθότι το θέμα είναι ένα θέμα με πολλές διαφορετικές πτυχές. Το θέμα των ε, οικονομικών υπηρεσιών, παραδείγματο χάρη. Δεύτερον, κοινωνικές υπηρεσίες. Κάτι που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Επίσης, η σχέση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών ε, υπηρεσιών. Το θέμα των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών επίσης που έτσι και αλλιώς δεν μπορούν επίσης να καλυφθούν από την οδηγία και θα πρέπει να δούμε εδώ τι η αλληλεπίδραση υπάρχει από νομικής απόψεως. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε ένα κείμενο μιας οδηγίας για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς το πεδίο εφαρμογής. Να μην ξέρουμε δηλαδή ποια οδηγία εφαρμόζεται σε ποια κατηγορία υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν αυτό να ξεκαθαριστεί με μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ακόμα έχουμε πολλή εργασία. Αναφερθήκατε επίσης στο άρθρο 2.5, 2.12, το 3.13 αυτό το προσθέτω εγώ, αλλά και κάποια άλλα που πρέπει σαφώς να ξανασυζητηθούν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα των δημόσιων ε, δημοπρασιών, το θέμα που αναφέρατε κι εσείς σε σχέση με το eBay. Οι καταναλωτές σε αυτή την περίπτωση, όταν πρόκειται για τέτοιου είδους ηλεκτρονικές ε, εμπορικές συναλλαγές, Ενώ ξέρουμε βεβαίως ότι δεν πρόκειται μόνο για πολίτες, για καταναλωτές, αλλά πολλές φορές αυτές τις ε, εμπορικές συναλλαγές λαμβάνουν χώρα και επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να μην ανοίξουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε και αυτές τις περιπτώσεις συμμετοχής. Και αυτό θα πρέπει κατά την άποψή μου να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε, αν και αυτό δεν επήγει τόσο, το θέμα των εμπορικών πρακτικών και ιδιαίτερα θα πρέπει να κοιτάξουμε πως κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν ανήκουν 100% στις οικονομικές υπηρεσίες, αλλά έχουν σχέση με την οδηγία για την πιστοτική πολιτική. Πρόκειται για τα ποσά αυτά που είναι κάτω από 75.000, ε, για την πιστοτική πολιτική η οποία θα πρέπει και εδώ να μπορεί να διασφαλίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, γιατί βλέπουμε πολλές φορές ότι ιδιαίτερα για τους νέους γίνονται προσφορές για δυνατότητα δανείων, ακόμα και με ένα απλό μήνυμα, ένα απλό SMS. Εδώ λοιπόν θα πρέπει πραγματικά να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα αυτών των νέων κυρίως καταναλωτών, αλλά πιστεύω ότι το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή και έχουμε αποφασίσει ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε ξεχωριστά. Παίζει όμως και αυτό το θέμα κάποιο ρόλο και έχει επιπτώσεις και θα πρέπει να το δούμε και σε σχέση με την οδηγία ή την προστασία των καταναλωτών. Τώρα το άρθρο 4. Δεν θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί ό,τι έχει σχέση με αυτό το άρθρο 4 έχει επίπτωση σε όλα τα άλλα άρθρα. Για μένα αυτό το θέμα θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε πρώτα. Θέλουμε εναρμόνιση ή δεν θέλουμε εναρμόνιση. Αυτό είναι το ερώτημα. Να σας διαβάσω το άρθρο 4. Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να διατηρήσουν στο εσωτερικό τους δίκαιο είτε να υιοθετήσουν οποιαδήποτε διάταξη η οποία δεν ε, συμβαδίζει με, ή αποκλίνει από αυτές τις διατάξεις. Το θέμα λοιπόν είναι εδώ αν λιγότερο αυστηρές διατάξεις στο εσωτερικό δίκαιο, στην εσωτερική νομοθεσία των κρατών, προστατεύουν εξίσου τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ να το αγνοήσουμε αυτό, γιατί μιλάμε εδώ για μια ελάχιστη εναρμόνιση, μια ελάχιστη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και το ερώτημα είναι Θέλουμε, ναι ή όχι, να το ξαναδούμε αυτό. Το θέμα της πλήρους εναρμόνισης, παραδείγματος χάριν, είναι ένα ερώτημα που τίθεται από την άλλη μεριά. Εάν δεν το ξεκαθαρίσουμε σε αυτήν την οδηγία, δεν θα το ξεκαθαρίσουμε ποτέ, διότι τα αγαθά, οι υπηρεσίες το βλέπουμε όταν συζητάμε τα θέματα στον τομέα των ε, τηλεπικοινωνιών. Κάθε φορά προκύπτει το ίδιο θέμα και τα δικαιώματα των καταναλωτών και η προστασία τους που κάθε φορά περνάνε μέσα από τα αιτήματα των ε, ενώσεων των καταναλωτών ε, λαμβάνουν απαντήσεις Τα κράτη-μέλη. Εάν θέλουμε εδώ εναρμόνιση θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή τη διαδικασία και αυτό το μηχανισμό. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Εγώ προσωπικά σας απαντώ όχι. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να ξανασυζητηθεί το θέμα αυτό στο κεφάλαιο 2, υποχρέωση ενημέρωσης και εδώ το θέμα της καταναλωτικής πίστης. Και εδώ δηλαδή υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης πληροφοριών Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς εδώ να μιλάει μόνο για την αντίδραση των ε, καταναλωτών και αν όντως λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις από τη στιγμή που δεν δίνονται οι σωστές πληροφορίες, δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Κεφάλαιο 3. Δικαίωμα και δυνατότητα επιστροφής ε, για περιπτώσεις ε, εμπορικών συναλλαγών που γίνονται στο σπίτι του καταναλωτή. Η δυνατότητα αυτή, το δικαίωμα αυτό εγγράφεται στην πρόταση και ιδιαίτερα όταν αναφέρομαι στις παραβιάσεις του άρθρου 9. Εδώ το δικαίωμα αυτό αναφέρεται για μία περίοδο που δεν ξεπερνάει τους τρει μήνες. Εδώ όμως θα υπάρχει πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, με το γερμανικό δίκαιο. Γιατί στη Γερμανία έχουμε μόνο ένα μήνα. Εάν όμως και εφόσον δίνονται όλες οι πληροφορίες. Εάν δεν είναι πλήρης οι πληροφορίες, θεωρείται ότι αυτό το δικαίωμα ουσιαστικά επιμικίνεται επάπειρον. Βλέπετε λοιπόν ότι παραδείγματο χάρη για τη Γερμανία περιορίζεται πάρα πολύ σημαντικά με αυτή τη νέα ε, πρόταση το δικαίωμα του καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε τι ακριβώς ε, συνέπειες έχει αυτό το άρθρο. Διότι δεν είναι μόνο θέμα προθεσμίας, γιατί ναι μεν ο ένας μήνας γίνεται τρεις, αλλά, αλλά από ποια στιγμή και πέρα αρχίζει να υπολογίζεται αυτή η προθοσμία Στην πράξη λοιπόν επιδεινώνεται η κατάσταση του καταναλωτή και δεν προστατεύονται εξίσου τα δικαιώματά του. Και υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα που θα μπορούσα να σας δώσω. Αλλά επειδή και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο, θα ξαναπάρω το λόγο ενδεχομένως αργότερα όταν ε, επεξεργαστούμε το θέμα αυτό και συζητήσουμε για τα υπόλοιπα άρθρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκέπχαρτ. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε πολύ περίπλοκες λεπτομέρειες. Όντως, χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Και νομίζω ότι ο εισηγητής, ο κ. Σφάμπ, έτσι και αλλιώς, το ανέφερε αυτό. Θα έχουμε όμως χρόνο να επανέλθουμε. Ο κύριος Ροσφό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ στον εισηγητή. Είμαστε σκιώδεις εισηγητές και τον ευχαριστώ πολύ γιατί μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε το θέμα εγκαίρως. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης γιατί νομίζω ότι όντως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να δούμε πιο ξεκάθαρα. Είπατε Επίσης, Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πρέπει, ποιοι είναι οι στόχοι. Ποιοι είναι οι καταρχήν της Επιτροπής και πώς μπορούμε να τους ιεραρχήσουμε. Πρώτον, απλοποίηση των κανόνων. Ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Τρίτον, να μειωθεί η αντίδραση των επιχειρήσεων όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο και θα προσθέσω και ένα τέταρτο στόχο, να υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο προσαρμόζεται σε έναν εξελισσόμενο κόσμο όπου τα προβλήματα της κατανάλωσης διαρκώς αλλάζουν. Και αν επιμένω σε αυτά τα τέσσερα σημεία, αυτό το κάνω γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα αξιολογηθεί η δράση μας όταν μεταφερθεί αυτή η οδηγία βάσει αυτών των στόχων. Εάν κάνουμε κάτι το οποίο περιπλέκει τα πράγματα και δεν τα απλοποιεί, δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή η οδηγία. Εάν δημιουργήσουμε περισσότερη δυσπιστία και όχι εμπιστοσύνη, επίσης. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είμαι πεπισμένος ότι για να υπάρξει σύγκληση θα πρέπει καταρχήν να προχωρήσουμε σε μια δράση που θα είναι χρήσιμη και για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σύγκληση και όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών και όσον αφορά τα δικαιώματα και τα ωφέλη των επιχειρήσεων. Για μια τόσο σημαντική οδηγία, οι επιπτώσεις για την καθημερινή ζωή είναι πολύ σημαντικές, για εκατομμύρια Ευρωπαίους που εκπροσωπούμε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να στηρίξουμε το τελικό κείμενο. Και αυτό γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρεία στήριξη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο χρόνο, καθότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, και συμφωνώ με τους δύο προηγούμενους ομιλητές, υπάρχει σήμερα αμφιβολία για πολλά σημεία, όπως και ο κύριος Φαμπ, έτσι ε, ακριβώς όπως έκανε και η κυρία Γκέπχαρτ, θα σας δώσω και εγώ για τα τρία αυτά κεφάλαια κάποια σημεία. Στο πρώτο κεφάλαιο, που αναφέρομαι στα πεδία εφαρμογή. πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να γίνει μια διασαφήνιση αυτών των πεδίων εφαρμογή. Συνάντησα ειδικού στον τομέα των ασφαλιών, οι οποίοι διαβάζοντας το κείμενο δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν, να καταλάβουν ποια τμήματα της δραστηριότητάς τους ενσωματώνονταν σε αυτή την οδηγία και ποια όχι. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν είναι ασαφές το πεδίο και αν ζητήσουμε πλήρη εναρμόνιση ή τη μέγιστη πιθανή εναρμόνιση, θα βρεθούμε διαρκώς μπροστά στα δικαστήρια και θα πρέπει να περιμένουμε κάθε φορά τη διαιτησία των δικαστών έτσι ώστε να βρεθεί το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εάν ε, υιοθετήσουμε την μέγιστη εναρμόνιση, δεν είναι δυνατόν να είναι ασαφές το πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλιώς δεν υπάρχει νομική ασφάλεια. Για το άρθρο 4 τώρα. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέει ο κύριος Φαμπ, ο οποίος λέει ότι πρέπει να το σκεφτούμε. Η κυρία Γκέπχαρ αντίθετα λέει ότι εάν δεν πάρουμε θέση όσον αφορά το 4, το όλο οικοδόμημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο. Εγώ βεβαίως και έχω πολλές επιφυλάξεις, αλλά το θεωρώ κρίμα να μην μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ελάχιστη εφαρμογή αυτής της μέγιστης εναρμόνισης. Τουλάχιστον μεταξύ μας θα πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτήν την μέγιστη εναρμόνιση και να συνειδητοποιήσουμε ότι εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία μέγιστη εναρμόνιση σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί οι περισσότεροι από εμά συνειδητοποιούν ότι δεν είναι δυνατόν να επιδεινωθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στα κράτη-μέλη. Και εάν οδηγηθούμε προς μία μέγιστη εναρμόνιση, δεν θα υπάρξει η απαραίτητη ευελιξία όσον αφορά το πεδίο της κατανάλωσης. Οι εθνικές ρυθμίσεις δηλαδή θα πρέπει να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν που υπάρχουν ε, σημεία στα οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί το κείμενο. Τώρα, εάν η μέγιστη ενερμόνιση είναι πολύ ευρεία, ενδεχομένως θα πλησιάσουμε έναν κανονισμό και δεν ξέρω αν σήμερα, στο επίπεδο που βρίσκεται η συνθήκη της Λισαβόνας, που ενδυναμώνει τα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σε λίγε μέρε θα υπάρξει ο διάλογος μεταξύ ημών και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ να πλησιάσουμε με ένα κανονισμό, να ζητήσουμε μια πολύ ευρεία εναρμόνιση, κάτι που θα δυσκολέψει αυτό το διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια. Για το άρθρο 4 λοιπόν σαφώς και θα πρέπει να επανέλθουμε γιατί είναι το κύριο θέμα. Όσον αφορά τον ορισμό που ανήκει επίσης στο κεφάλαιο 1, εγώ όσον αφορά τον ορισμό του καταναλωτή τον ορισμό που έχουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ περιοριστικός αυτός ο ορισμός και αναρωτιέμαι μήπως θα πρέπει να διευρυνθεί αυτός ο ορισμός έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και εμπορικές συναλλαγές οι οποίες ουσιαστικά έχουν σκόπο επαγγελματικό αλλά και ιδιωτικό. Όσον αφορά τώρα το κεφάλαιο 2, την ενημέρωση των καταναλωτών, εδώ δυσκολεύομαι ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή της μέγιστης εναρμόνισης σε ένα πεδίο το οποίο καλύπτει τόσους πολλούς τομείς, όπως προτείνει το κείμενο. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έναν κατάλογο πλήρη για όλους τους τομείς. Και θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δύο κατηγορίες υπηρεσιών. Την κομμωτική από τη μία και τους οίκους ευγυρίας. Υπηρεσίες που πολλές φορές όσον αφορά τους οίκους ευγυρίας αναφέρονται σε ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών. Πώς μπορούμε λοιπόν εδώ να καθορίσουμε ενημέρωση που να είναι ταυτόσιμη για αυτούς τους δύο συγκεκριμένους κλάδους. Και αυτό βεβαίως ισχύει και για πάρα, πολλά άλλα, ε, πάρα πολλές άλλες κατηγορίες υπηρεσιών. Για το κεφάλαιο 3, επίσης, το άρθρο 9, 10 και 11, που εξαρτώνται από το άρθρο 5 όσον αφορά την εξαποστάσεως πώληση, παραδείγματος χάρη, και όπως σήμερα καθορίζονται αυτά τα άρθρα, υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία που οι διατάξεις σήμερα είναι πιο αυστηρές και προστατεύουν περισσότερο τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να συνεχίσουμε τη συζήτηση για όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να βρεθεί η διαδικασία βελτίωσης του κειμένου. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι η μέγιστη αναρμόνιση παρόλα αυτά θα μπορούσε να εφαρμοστεί για όλα τα άρθρα που ακολουθούν το άρθρο 11. Ιδιαίτερα όσον αφορά την προθεσμία για την επιστροφή της εξαιρέσεις και τα λοιπά. Πολύ λοιπόν εργασία ακόμα πρέπει να γίνει. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί επιτέλους μπήκαμε στην ουσία του θέματος. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε την εργασία μας και επί των αρχών και επί της εφαρμογής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ροσφόρ για τη συνεισφορά σας. Νομίζω ότι συνοψίσατε πολύ κομψά όταν είπατε ότι εδώ προσπαθούμε να έχουμε τελέξει τα επιτεύγματα της μέχρι της Έτσι λοιπόν κατανοούμε τι είδους προβλήματα έχουμε προς στιγμή. Η κυρία Τούνα και ο κύριος Τριανταφυλλίδης ε, και ο κύριος Μπίλεν δεν ξέρω αν θέλει να συνεισφέρει. Και να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι πρέπει να ξεκινήσουμε στις 4.30 την ακρόση, γιατί θα έχουμε πολλούς ε, ομιλητές. Νομίζω ότι βέβαια θα υπάρχουν και πολλές ε, ευκαιρίες ε, για την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σφαπ. Δεν θέλω να σας βιάσω, απλώς να σας πω ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Κυρία να ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον συζητητή που έλαβε το χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και δεύτερον ε, εκτιμώ την προθυμία του να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι είναι καλή αφετηρία. Για το κεφάλαιο 1-3 νομίζω ότι αυτό αυτό είναι το πιο εύκολο τμήμα της οδηγία, ε, αλλά αυτό είναι και το πιο δύσκολο, γιατί ουσιαστικά θα το σκηνικό για τα υπόλοιπα. Σήμερα δεν θα σχολιάσω λεπτομερώ επί των άρθρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση, αλλά θα ήθελα να εξάγω κάποια συμπεράσματα γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στο background, ε, στα μοτίβα και στη βάση των πληροφοριών ε, και δεν νομίζω ότι πρέπει να τα παραβλέψουμε αυτά. Καλωσορίζουμε λοιπόν ε, αυτή την οδηγία και υποστηρίζουμε την ε, κατεύθυνση, αυτό αναφέρθηκε και από άλλους, στο να συνεισφέρει στην ε, καλή λειτουργία της ενής αγοράς και να πετύχουμε ύψιστη προσδεσία του κανόνων. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά, αλλά πιστεύουμε ότι η οδηγία δεν είναι ολοκληρωμένη ως προς το εργασίες που έχουν γίνει. κατά την ε, διάρκεια της σύνταξης, εμείς θεωρούμε ότι έχουν ε, αγνοηθεί οι απόψεις των ενδιαφερόμενων περών. Εμάς μας ε, ενδιαφέρει τι γίνεται με την εναρμόνιση, γιατί είναι ασαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους κανονιστές σε κάθε κράτος μέλος. Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία, καμία αρχή κράτος μέλος που μπορεί να δω, κάνει μία ε, ακριβή αξιολόγηση των νομικών συνεπειών. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ανησυχία και νομίζω ότι είναι ανησυχητικό ότι στα κράτη-μέλη, στα όλα τα κράτη-μέλη, οι νομικοί έχουν δυσκολίε να κατανοήσουν πώς η κοινωτική νομοθεσία και η εθνική νομοθεσία θα συντεριάξουν. Ε, εμεί είδαμε και μία μελέτη που υλοποίησε ο κ. Χάνσον Κινούλκιν ε, από το Πανεπιστήμιο του Χάντσεμπουργκ ελοποίησε μία μελέτη για την Επιτροπή Γιούρη και θα σας πω ότι είπε ότι η προσέγγιση της πρότασης μπορεί να έχει επιπτώσει σε πολλά κράτη-μέλη και να οδηγήσει σε παράδοξες καταστάσεις. Αν ε, ε, οι καταναλωτές περιοριστούν στα ένδικα μέσα που προτείνονται, τότε θα βρίσκονται σε χειρότερη θέση από ότι μη καταναλωτές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που λέγεται εδώ. Εμείς ε, προτείνουμε ότι σε, ορισμένες, σε ορισμένους ορισμούς, παραδείγματος χάρη, η πλήρης εναρμόνιση θα μπορούσε να έχει νόημα, αλλά έχουμε πάρα πολύ λίγη εμπειρία με την πλήρη εναρμόνιση σε αυτό το τομέα και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ζητάμε περισσότερε πληροφορίε και να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στι νομικέ επιπτώσει που θα υπάρχουν στα κράτη-μέλη αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο πριν να συνεχίσουμε το εγχείρημα. Ακόμη, να πω και κάτι σε ό,τι αφορά το background. Δηλαδή αναφέρθηκε το θέμα της αύξησης του διασυνορικού εμπορίου, ότι αυτός είναι ένας λόγος ε, για την εκπόνηση της νομοθεσίας, όμως η έλλειψη της εναρμόνισης δεν είναι ε, το κύριο πρόβλημα που έχουμε αν δούμε τις διασυνορικές συναλλαγές. το χάρη, σύμφωνα με στοιχεία του 2008, το 70% των εταιριών είπαν ότι αυξημένη εναρμόνιση δεν θα έχει, έχει πολύ λίγη επίπτωση στις διασυνοριακές πωλήσει. Δεν υπάρχουν λοιπόν αποδείξεις για το πώς ε, αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών η οδηγία και πώς προωθεί το διασυνοριακό εμπόριο. Το περιεχόμενο της οδηγία φαίνεται να βασίζονται στην ε, υπόθεση και σε, υπερ, σε μια υπόθεση σε υπερεκτίμηση ε, των ε, εμποδίων που υπάρχουν στο διασυνοριακό εμπόριο. Όμως εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα συνοψίσω λοιπόν κάποια συμπεράσματα. Φυσικά αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα ε, να υπάρχει μια νομοθεσία που να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και των αγορών, αλλά είμαστε πολύ σκεπτικοί απέναντι ε, στην προσέγγιση της Κομισιόν. Να σα πω και το εξή. Δεν είναι καλά προετοιμασμένη η οδηγία, δεν έχουμε επαρκεί προφορίε για τον αντίκτυπο. Ανησυχούμε ότι η πλήρη εναρμόνιση αυτή η στρατηγική όπω προτείνει την Κομισιόν θα αποδυναμώσει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Πρέπει να μην αποδυναμωθούν από αυτή την οδηγία τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι ε, τελικά θα ευνοηθεί το διασυνοριακτό εμπόριο, όπως προτείνεται. Βέβαια, να το διαρευνήσουμε. Είμαστε πρόθυμοι. Και τέταρτο, για αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να συστήσουμε τη συνέχιση της διαδικασίας ε, πριν έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Έτσι, λοιπόν, εμείς ως Επιτροπή πρέπει να συνεχίσουμε να ζητάμε περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες επί, της, ε, επί των οποίων θα εκπονήσουμε νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να συνεχίσουμε χωρίς να γνωρίζουμε επί ποιου πράγματος συντάσσουμε νομοθεσία και ποιε είναι οι συνέπειε. Έτσι λοιπόν, σα ενθαρρύνω όλου να συνεχίσετε να ζητάτε αυτή την ενημέρωση για την περαιτέρω διαδικασία, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή βάση για να χτίσουμε την νομοθεσία μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σαφή σα σχόλια για τη στρατηγική προσέγγιση. Είναι σχόλια εκ μέρου της Επιτροπής ότι φυσικά αυτή τη διαδικασία ε, της συλλογή πληροφοριών την ξεκινήσαμε 6 μήνες πριν από τι εκλογές και μπορείτε να δείτε και την έκθεση εργασία τη κυρία Μακαρθ. Υπάρχουν κάποιε πληροφορίε. Και έτσι λοιπόν η γραμματεία έχει πάρα πολλά δεδομένα ε, που τα έχει συλλέξει και δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις ε, και φυσικά αν συνεχίσουμε να ζητάμε περισσότερε πληροφορίε προς την κατεύθυνση που ζητήσετε θα συνεχίσει να το πράττει ο συγητής, ο κ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Άντρια ε, ε, Σβάπ για την πολύ ωραία και καταδεκτική στάση που τηρεί αντί όλων των πολιτικών ομάδων. Έχει ακούσει και εμά και ε, είμαι σίγουρο ότι οι απόψει που εκφράστηκαν θα ληφθούν υπόψη. Σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω στα πρώτα τρία κεφάλαια, όπως είναι και η εισήγηση του εισηγητή, και να περιοριστώ στα σημεία πάνω στα οποία ε, εντοπίζουμε κάποιες ε, διαφορές για να βοηθήσουμε ίσως την εξέβρεση μιας κοινή συνισταμένης. Στο κεφάλαιο 1, που αφορά τους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής, θα αναφέρω τρία σημεία τα οποία πρέπει να προσεχτούν. Έχουμε την εντύπωση ότι η πλήρης εναρμόνιση ισοδυναμεί με ξεκάθαρη μείωση της προστασίας των καταναλωτών ότι αφαιρεί από τα κράτη-μέλη ε, τη δυνατότητα να λαμβάνουμε μέτρα που ανταποκρίνονται στις αντικειμενικές συνθήκες της κάθε χώρας. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά τις εγγύησεις στο τέταρτο κεφάλαιο, μειώνει το εφιστάμενο πεδίο προστασίας των καταναλωτών στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τη μελέτη που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα κράτη-μέλη. Και ήθελα να σημειώσω επίσης ότι με την εφαρμογή της πλήρους εναρμόνισης αυτοί που επωφελούνται κυρίως από τη μείωση των διοικητικών κόστων είναι οπωσδήποτε οι επιχειρήσεις χωρίς η μείωση αυτή να φαίνεται να συνδέεται σε κανένα σημείο της οδηγίας με μείωση του κόστους για τους καταναλωτές. Στο κεφάλαιο 2 που αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών μας ανησυχεί το σημείο που αφορά στην πληροφόρηση για τις τιμές Έχουμε τη γνώμη ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει την τιμή και τις επιπρόσθετες επιβαρύνσεις σε κάθε περίπτωση. Ότι οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται αναλυτικά σε κάθε περίπτωση για να μην παραπλανούνται οι καταναλωτές ως προς το τελικό κόστος του προϊόντος. Στο κεφάλαιο 3, που αφορά την περίοδο υπαναχώρησης για τις εξαποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις εκτός καταστήματος, διαφωνούμε με την πρόνοια στο άρθρο 14 που υποχρεώνει τον καταναλωτή να ενημερώνει για την επιθυμία του να υπαναχωρεί, γιατί αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία περιορίζει οπωσδήποτε τη δυνατότητά του να υπαναχωρεί. Και επίσης το άρθρο 12, σχετικά με την αφετηρία της περίοδου υπαναχώρησης, πιστεύουμε ότι η περίοδος μέχρι την παράδοση του προϊόντος δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην περίοδο υπαναχώρησης. Άρα η έναρξη της περίοδου υπαναχώρησης θα πρέπει να τίθεται σε ισχύ από την παράδοση του προϊόντος και όχι από την παραλαβή του εντύπου παραγγελίας. Και τελειώνοντας ήθελα να πω ότι η γενική εντύπωση που παίρνουμε είναι ότι το περιεχόμενο της οδηγίας δεν συνάδει με τον τίτλο της. Δηλαδή η προστασία των καταναλωτών περιορίζεται στο βαθμό που αυτή δεν επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν προϋποθέτει επιπλέον κόστος για αυτές. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την αρχή και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημαντικές ευθύνες να διασφαλίσει την παροχή υψηλού επίπεδου προστασίας των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τριανταφυλλίδη και κύριε Κράτσπιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατανοώ τι ανησυχίε ε, των συναδέλφων και κυρίω ε, του ηγητή κ. Βαμπ για το ότι είναι πολύ πλόκο το θέμα και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Όμω, για την πλήρη εναρμόνιση, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να μην μειώσουμε τα πρότυπα τώρα. Πρέπει ουσιαστικά να διατηρήσουμε τον έσχατο στόχο που έχουμε για πλήρη εναρμόνιση και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα βήμα το βήμα ρεαλιστικά. Πρόβλημα το πρόβλημα. Σε ξεχνάμε ότι η εναρμόνιση αυξάνει τον ανταγωνισμό και διευκολύνει το εμπόριο και μας δίνει μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν όλοι και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Τώρα, εγώ μιλώ γιατί έχω άμεση εμπειρία, επειδή ε, γνωρίζω πώς ε, κάποιος πρέπει να διευθύνει μια μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη και εγώ νομίζω ότι πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτό γίνεται με σαφήνεια και φυσικά για μια εταιρεία μικρή είναι σαφές ότι και για μένα και για πολλούς άλλου που διευθύνουν μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη, η κατακαιρμάτιση τη νομοθεσία είναι κόστο και είναι διοικητικό άχθο. Να πω και στη δράση συνάδελφο ότι συμμερίζομαι τι ανησυχίε τη. η Σουηδία η οποία έχει πολύ ψηλά πρότυπα Προστασία του καταναλωτή είναι έτοιμη να ε, εγκαταλείψει μερικά. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για εγκαταλείψη εδώ, απλώς θεωρούμε ότι η πλήρη εναρμόνιση θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Και αν έχετε μία νομοθεσία που να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης ε, θα μπορέσετε να έχετε και εκστρατείε ενημέρωσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσει. Ναι, περισσότερος χρόνος, ναι, τι πληροφορίε, αλλά είμαστε εδώ για να παράγουμε αποτελέσματα και ελπίζω αυτό να μην γίνει σε δύο χρόνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για τις ε, ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους που νομίζω θα είναι χρήσιμες για τον εισηγητή. Θα ήθελα να καλέσω τον Τζάκη Μάινερ από την Επιτροπή να ε, σχολιάσει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, θα υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες να μιλήσει, αλλά δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει και κατόπιν θα ζητήσω από τον Άντρου Σφάπ να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη. Κάποιες προκαταρτικές παρατηρήσεις. Δεν θα σας κουράσω με αυτά που είπα στην προηγούμενη συνεδρία, αλλά θα, θα ήθελα να συμφωνήσω με την τελευταία ομιλήτρια. Η πλήρης εναρμόνιση αποτελεί κατάσταση από την οποία θα κερδίσουν όλοι. Ο κύριος Ροσφόρ συνόψισε πολύ σωστά την κατάσταση και πιστεύουμε ότι υπό το φως αυτό η πλήρης εναρμόνιση είναι η μόνο προσέγγιση που ε, θα δώσει στις επιχειρήσεις μια σειρά από απλούς ε, κανόνες ε, σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να εργάζονται και εξασφαλίζει για τους καταναλωτές το ίδιο επίπεδο προστασίας όπου και αν αγοράζουν κάτι, είτε αγοράζουν κάτι σε ένα κανονικό μαγαζί, είτε επιγραμμικά μέσω ίντερνετ. Η κυρία Τούρινεν παρέθεσε κάποια λόγια του καθηγητή ο οποίο ε, αμφισβητεί την πλήρη εναρμόνιση. Νομίζω όμως ότι ε, παρέθεσε τα λόγια αυτά έξω από το περιβάλλον τους, διότι αναφέρεται στην εξαντλητική πλήρη εναρμόνιση και όχι τη στοχευμένη εναρμόνιση που προτείνει η Επιτροπή. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την αύξηση ή μείωση του επίπεδου προστασίας. Αυτό συζητιέται από όλους τους ενδιαφερόμενους. Συζητήθηκε και πριν υποβληθεί η πρόταση και συνεχίζει να συζητιέται. Η συνθήκη μας αναγκάζει να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Και συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι το επίπεδο προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα αυξηθεί με την πρόταση αυτό. Βέβαια, είναι εξίσου αλήθεια ότι το αποτέλεσμα της πλήρους εναρμόνισης είναι ότι κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να τροποποιήσουν κάποιες πτυχές της ε, ισχύουσας ε, ε, νομοθεσίας τους για τον καταναλωτή. Αλλά το επίπεδο στο σύνολο των 27 κρατών μελών θα αυξηθεί. Η Επίτροπος έχει επανειλημμένα πει και το είπε και τελευταία φορά στην Επιτροπή σας. ότι θέλουμε κατάλληλο επίπεδο εναρμόνισης. Δεδομένης της πολυπλοκότητας, ε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι είναι όντως μια πολύπλοκη πρόταση, ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι η πρόταση αυτή έχει περάσει από εξαντλητική διαδικασία διαβούλευσης, πολύ προσεκτική αξιολόγηση και πιο ασυνήθιστο είναι ότι έχει συζητηθεί, έχει ερμηνευθεί ή έχει εξηγηθεί από το, την Επιτροπή. έχει ε, εξεταστεί για παράδειγμα ο βαθμός στον οποίο η πρόταση αυτή ε, θα επηρεάσει την νομοθεσία των ε, κρατών μελών, κάτι που συνήθως αξιολογούν τα κράτη-μέλη στη διαδικασία εφαρμογής, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η Κομισιόν εκπώνησε ένα κατάλογο. Μάλιστα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προσπάθησαν να εξετάσουν τις επιπτώσεις στην εθνική νομοθεσία πριν την ε, υιοθέτηση από το Συμβούλιο. Ε, αυτό έγινε δεδομένη της πολυπλοκότητα της πρότασης. Όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο και την προώθησή του. Εδώ φοβάμαι θα πρέπει να διαφωνήσω. Στην ε, μελέτη επιπτώσεων αναφέρουμε ε, στοιχεία από το ε, μελέτη του Ευρωβαρόμετρου του 2008. Δεχόμαστε ότι ο νομικός κατακαιρματισμός, δεδομένου το ότι υπάρχουν 27 διαφορετικά ε, νομικά καθεστώτα για τις συμβάσεις των καταναλωτών, δεν είναι το μόνο εμπόδιο στο διασυνοριακό εμπόριο. Και η γλώσσα και η κουλτούρα της κάθε χώρας είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες. Ω νομοθέτες όμως πιστεύουμε ότι ο νομικό κατακαιρματισμό αποτελεί σημαντικό αντικίνητρο για τους εμπόρους που αλλιώς θα πουλούσαν σε καταναλωτές στα άλλα κράτη-μέλη. Το 2008 από τους εμπόρους που δεν πολλούν σε άλλο κράτος μέλος 70 5% όλων των επιχειρήσεων, η μισοί από αυτούς είπαν ότι θα το έκαναν εάν υπήρχε εναρμόνιση των κανόνων. Αυτοί λοιπόν που, από του, αυτούς που δεν το κάνουν αυτή τη στιγμή, οι μισοί τουλάχιστον, θα ενθαρρύνονταν να απολούν σε καταναλωτές σε άλλα κράτη-μέλη εάν πετυχαίναμε εναρμόνιση της νομοθεσίας. Και σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώσαμε ότι πάνω από 6 από 10 συναλλαγές που προσπάθησαν να κάνουν καταναλωτές απέτυχαν επειδή οι επιχειρήσεις αρνήθηκαν να πουλήσουν διασυνοριακά. Υπάρχει λοιπόν ευκαιρία να βρουν επιχειρήσεις νέους πελάτες, υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες για τους καταναλωτές, διότι η ίδια μελέτη έδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις Ακόμα και αν, ε, αυξήσει κανείς, ε, ακόμα και αν προσθέσει κανείς ε, έξοδα αποστολής, ο καταναλωτή μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα αγοράζοντας κάτι από άλλο κράτο μέλο. Πολύ σύντομα ε, να κάνω κάποιες πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις ε, όσον αφορά αυτά που είπε ο εισηγητής και άλλοι. Αναγνωρίζω την ε, δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά τη συμπερίληψη των υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι νέο. Οι υπηρεσίες ήδη συμπεριλαμβάνονται στην ε, οδηγία για τις αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ ε, και για τις πωλήσει εκτός εμπορικού καταστήματος. Ε, πρόκειται λοιπόν για ενοποίηση του καταναλωτικού κεκτημένου και βλέπουμε και στις υποθέσεις του δικαστηρίου ότι τα, οι διασυνοριακές συμβάσεις, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, είναι πολύ συνηθισμένες. Εάν αφαιρέσουμε λοιπόν τις υπηρεσίες στο σύνολό τους, αυτό θα υπονομεύσει το, τον αντίκτυπο της πρότασης. Όσον αφορά το ορισμό του προϊόντος στο άρθρο 2 σημείο 12 είναι ο ίδιος ε, με, την, ε, με αυτόν που υπάρχει στην ε, οδηγία για τις αναθέτητες εμπορικές πρακτικές. Βασιζόμαστε δηλαδή στο κεκτημένο. Επίσης, οι δημοπρασίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Σφάπ και η κυρία Κέπχαρτ. Αυτό είναι δύσκολο ζήτημα. Ξέρω ότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ε, απόψεις σχετικά με το τι είναι δίκαιο και τι όχι και το ποιο θα πρέπει να προστατευτεί. Θα πρέπει να προστατευτεί ο υπερθεματιστής ή θα πρέπει να προστατευτεί ή θα πρέπει να προστατευτούν οι καταναλωτές οι οποίοι τελικά δεν κερδίζουν στη δημοπρασία και που μπορεί τελικά ε, εάν αποσυρθεί ο υπερθεματιστής ε, να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Όσον αφορά την ενημέρωση, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Συμφωνούμε ότι οι υπερβολικά πολλές πληροφορίες ε, δεν βοηθάνε. Σημειώνω τις ανησυχίε του ε, εισηγητή σχετικά με τις εφημερίδες που απολούνται εκτός εμπορικού καταστήματος. Ο συνάδελφός μου θα αναφερθεί στο ε, πολύπλοκο ζήτημα των ε, ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και ξέρω ότι στη Γερμανία και στην Αυστρία όταν ε, δεν λαμβάνει κανείς επαρκή πληροφορία σχετικά με το δικαίωμα επαναχώρηση, ο χρόνος δεν ξεκινάει να τρέχει για τον καταναλωτή, παρά μόνο όταν διορθωθεί η κατάσταση. Ε, αυτή δεν είναι η επιλογή που ζητήσαμε, ε, η επιλογή που επιλέξαμε σε αυτή την πρόταση, ούτε στην ε, οδηγία της χρονομεστικές μισθώσεις. Θέλουμε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα του εμπόρου και στα δικαιώματα του καταναλωτή. Και πιστεύουμε ότι η λύση μας ε, παρέχει μεγαλύτερο βαθμό ασφαλείας δικαίου. Το άρθρο 13 αναφέρεται αποκλειστικά στο δικαίωμα υπαναχώρησης ε, και όχι στα άλλα ένδικα μέσα ε, στα οποία μπορεί να προσφύγει ο καταναλωτής. Όσον αφορά τον ορισμό του καταναλωτή, Ισχύει αυτό και για προϊόντα που προορίζονται εν μέρη για ε, επαγγελματικούς σκοπούς και εδώ έχουμε βασιστεί στην υπάρχουσα πρακτική. Εξετάζουμε δηλαδή τον κύριο λόγο για τον οποίο αγοράζονται τα προϊόντα. Πιστεύουμε ότι έτσι πετυχαίνουμε τη σωστή ισορροπία όσον αφορά την ισορροπία ανάμεσα στον καταναλωτή και τι επιχειρήσεις. Τέλος, απαντώντα στον κύριο Τριανταφυλλίδη, το θέμα της υπαναχώρηση. Πότε ξεκινάει η προθεσμία. Γίνεται διάκριση ανάμεσα στις ε, συμβάσεις εξ αποστάσεως και στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος για τις ε, συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος ε, οι δύο εβδομάδες ξεκινάνε από την υπογραφή του εντύπου παραγγελίας. Κανονικά σε ε, συμβάσει εκτός εμπορικού καταστήματος ο καταναλωτής έχει κάποια ιδέα για το τι αγοράζει. Έχει τη είχε τη δυνατότητα να το εξετάσει αυτό το θέμα, είναι να τον προστατεύσουμε από την ψυχολογική πίεση που προκύπτει όταν ο πολιτής βρίσκεται στο σπίτι του καταναλωτή ή εκτός εμπορικού καταστήματος. Για τις άλλες συμβάσεις η προθεσμία ε, ξεκινάει από την παραλαβή των προϊόντων από τον καταναλωτή. Θα σταματήσω εδώ και θα παρακαλέσω τον Ζουζέπε να απαντήσει σύντομα ε, στο θέμα των ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πρόεδρος, συγγνώμη Τζάκη. Νομίζω ότι μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Λυπάμαι πολύ. Απλά έχουμε άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αν μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας ε, γραπτό στον Άντριου Σφάρπ, ε, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Άλλωστε θα ακολουθήσει άλλη μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Θέλετε να πείτε κάτι ή μπορώ να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Χαιρόμαστε πολύ που είναι το Συμβούλιο εδώ και παρακολουθεί τις εργασίες μας. Άντριου, θες να συνοψίσεις πολύ σύντομα πριν κλείσουμε το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους και συγγητέ, ε, το Συμβούλιο, την Επιτροπή για, τις τους, ε, για την επικοδομητική τους ε, συμβολή. Ε, όποιος θέλει να υποβάλει προτάσεις, πολύ θα χαρώ να λάβω τις προτάσεις σας. Στη συζήτηση αυτή κανένας δεν είπε ότι α, στην πατρίδα μου κάνουμε έτσι και γι' αυτό δεν γίνεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό στην Ευρώπη. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοδομητικά ε, εξετάζεται τι γίνεται στα 27 κράτη-μέλη για να πετύχουμε ε, ένα υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών. Και φυσικά πιστεύω ότι οι επικρίσεις που ακούστηκαν ε, όσον αφορά την πλήρη εναρμόνιση είναι εν μέρη ε, δικαιολογημένες, αλλά μπορεί να διαπιστώσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η πλήρης εναρμόνιση όπως ε, υπάρχει στην πρόταση της Κομισιόν δεν μπορεί να επιτευχθεί και γι' αυτό είναι ενδιαφέρον ότι εδώ μπορούμε να συζητάμε τα διάφορα ζητήματα. Ελπίζω να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι και εγώ φυσικά ε, είμαι υπέρ της εσωτερικής αγοράς και ελπίζω με την ε, έκθεσή μου να μπορέσω να συμβάλλω στην καλύτερη λειτουργία της. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία σε ευχαριστήσω, Άντριου, ε, που ανέλαβε τον ηγετικό ρόλο και νομίζω ότι όλοι έχουν συνεισφέρει. Είναι σίγουρα η πιο σημαντική πρόταση που θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον και πρέπει να την εξετάζουμε με προσοχή. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ για την ακρόαση που θα έχουμε με το Γαλλικό Εθνικό Κοινοβούλιο και φυσικά θα έχουμε περαιτέρω ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει Ζητώ συγγνώμη από την Κομισιόν που δεν ε, την άφησα να ολοκληρώσει τα σχολεία της, ε, αλλά έχουμε και κάποια ακόμη θέματα και πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Σε ευχαριστώ όλους λοιπόν. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ό,τι αφορά το scoreboard των ε, καταναλωτικών αγορών. Χαίρομαι που ήρθατε, ε, γιατί νομίζω ήσασταν άρρωστοι. σε σχέση με τους πιο εισηγητές, κύριο Ρουσφόρ και εγώ είμαστε οι μόνοι που είμαστε εδώ από τους και οδησηγητές. Έτσι λοιπόν, αν συμφωνεί ο κύριος θα προτείνω στην περίπτωση αυτή, αν μπορούσατε να παρουσιάσετε το θέμα και τα κύρια θέματα και να μας πείτε ποιο είναι και το χρονοδιάγραμμα. Και στις 2 Δεκεμβρίου, στην επόμενη συνάντησή μας, θα κανονίσουμε πότε θα έχουμε μία πλήρη συζήτηση μαζί σας, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα την ακρόαση σε λίγο. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο και αν και ο κύριος Μαερ ε, θέλει να κάνει πιο σχόλιο, αυτό θα κάνουμε, αλλά να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφε. Πάντα ε, έλεγα ότι στην Επιτροπή μας ότι χρειαζόμαστε ικανοποιημένους ε, και ασφαλείς καταναλωτές για να μπορέσει να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Και ο καταναλωτής, ε, ο, ο πολίτης ως καταναλωτής ε, έχει την εμπειρία της εσωτερικής αγοράς στην καθημερινή του ζωή. Και γι' αυτό θα πρέπει να εργαζόμαστε συνέχεια ώστε να βρίσκουμε νέους τρόπους να ενισχύσουμε τα ε, δικαιώματα των καταναλωτών. Υπάρχει λόγος ε, να θεωρούμε ότι οι, εσωτερικοί, οι καταναλωτές ε, δεν απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ένα scoreboard, έναν πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές για την προστασία των καταναλωτών. Θα θυμάστε την πρώτη μας συζήτηση ε, του πίνακα αποτελεσμάτων. Ε, σχεδόν ε, ακριβώς πριν ένα χρόνο το Κοινοβούλιο άρχισε να ασχολείται με το θέμα. Μιλήσαμε για τους δείκτες τιμών και συμφωνήσαμε ότι η τιμή είναι μόνο ένας παράγοντας για να ε, αξιολογήσουμε την ε, λειτουργία της ε, αγοράς. Στις 28 Ιανουαρίου φέτος η Κομισιόν παρουσίασε τη δεύτερη εκδοχή του πίνακα αποτελεσμάτων και πάλι έγινε ανάλυση των καταναλωτικών αγορών με βάση τα ίδια κριτήρια που είχαμε στην πρώτη εκδοχή. Κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα ήταν ε, ότι οι καταναλωτές γενικά είναι λιγότερο ικανοποιημένοι ε, από τις υπηρεσίες από, ότι, από τα αγαθά. Κυρίως ε, όσον αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και τις τραπεζικές υπηρεσίες. Οι τιμέ είναι πιο χαμηλές στο τομεί όπου οι καταναλωτές συχνά αλλάζουν πάροχο. Σημαντικό λοιπόν είναι να μπορούμε να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητα και οι αγορές να είναι προσανατολισμένες στον καταναλωτή, διότι ο μη ικανοποιημένος καταναλωτής είναι πιο λογικό να αλλάξει πάροχο. Σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης είναι επίσης ότι οι διασυνοριακές ε, ηλεκτρονικές αγορές δεν έχουν αυξηθεί εξίσου με τις εθνικές. Μόνο 7% ε, των πολιτών αγοράζουν διασυνοριακά και το νούμερο αυτό είναι πολύ χαμηλό ο πίνακα ε, αποτελεσμάτων ε, είναι ακόμα νέος, είναι ένα μωρό το οποίο ελπίζουμε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ε, σιγά σιγά και θα πρέπει να έχουμε υπομονή και να έχουμε κάποια πράγματα κατά νου όταν εξετάζουμε τα αποτελέσματα αυτά. Για παράδειγμα δεν έχουμε τις ποιοτικές τα ποιοτικά δεδομένα που θα θέλαμε. Πολλά κράτη-μέλη δυσκολεύονται να συλλέξουν τα στοιχεία και ε, δεν ε, έχουν ακόμα καταφέρει να παρουσιάσουν τα δεδομένα αυτά στο ευρύ κοινό, διότι θέλουμε και ο απλός καταναλωτής να γνωρίζει τα στοιχεία αυτά. Κάτι που έχει αλλάξει από πέρσι είναι ότι έχουμε αλλάξει τον τίτλο της μελέτης. Ε, τώρα αναφερόμαστε στην προστασία του καταναλωτή. Έχουμε εξετάσει τις ε, προτάσεις ε, της Κομισιόν και έτσι μπορέσαμε να διευρύνουμε το πεδίο της έκθεσης αυτής, αν και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στον πίνακα αποτελεσμάτων και θα πρέπει να αποφύγουμε να εξετάζουμε τομείς που εξετάζονται σε άλλες εκθέσεις. Ωστόσο, υπάρχει λόγος να εξετάσουμε την, ε, τον κανονισμό για την συνεργασία στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τους σκιώδεις συζητητέ και τους συναδέλφους και στην συνέχιση της συζήτησης στις 2 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω ότι ίσως η 1η Δεκεμβρίου είναι καλύτερη ημερομηνία για να συνεχιστεί η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, 1 και 2 Δεκεμβρίου θα έχετε αρκετό χρόνο. Κύριε Ροσφόρ, συμφωνείτε. Θέλετε να σχολιάσετε, κύριε Μάρτ. Ναι, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι η Επιτροπή αποφάσισε να προετοιμάσει μια έκθεση. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα που σαφώς και κατέχει πολύ σημαντική θέση στις κατευθυντήριες γραμμές που προετοιμάζουμε. «27», κανάλι 27, για τα γερμανικά. Όπως έλεγα, Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η Επιτροπή αποφάσισε να προετοιμάσει μια έκθεση για το θέμα αυτό. Εάν ε, εξετάσετε τις κατευθυντήριες γραμμές του Πρόεδρου Μπαρόζο, θα δείτε ότι όντως το θέμα αυτό των μετρήσεων, των δικτών και της ε, επιτήρησης αγοράς παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο νέο πρόγραμμα με ένα συστηματικό τρόπο θέλουμε να παίξουμε αυτό το ρόλο στην αγορά. Να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η εσωτερική αγορά και ποιες είναι οι δυνατότητες βελτίωσης ικανοποίησης των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αυτός λοιπόν ο πίνακας με τους δείκτες και τις μετρήσεις είναι ένα πάρα πολύ ε, χρήσιμο εργαλείο για μας, όπως είπε και η συγγήτρια και πιστεύω ότι θα προοδεύσουμε πολύ σημαντικά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκδοχής. Ελπίζω ε, ότι η πρόοδος αυτή θα συνεχιστεί και σε κάποια μελλοντικά στάδια της εργασίας μας θα σας δώσουμε και κάποιες ημερομηνίες, προθεσμίες για το τι θέλουμε να κάνουμε το επόμενο έτος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία. Πιστεύω ότι η πρόταση της εισηγήτριας όσον αφορά τη διεύρυνση των προτάσεων ε, για να συμπεριληφθούν και κάποιες ε, δυνατότητες συμμετοχής των καταναλωτών είναι κάτι πολύ υλικό και το υποστηρίζουμε. Δεύτερον, αυτό είναι το έγγραφο για το οποίο συζητούμε. Ελπίζω να το έχετε όλοι. Ελπίζω να υπάρχει και η γλώσσα όλων σας, σε αυτό το έντυπο. Η συγγήτρια λοιπόν θα συνεχίσει την εργασία και ελπίζω την επόμενη φορά να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο λεπτομερή συζήτηση. Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά, κατόπιν θα αναλάβει η Αντιπρόεδρος ε, την ε, Προεδρία για την ακρόαση και θα καλέσω βεβαίως και όλους τους εμπειρογνώμονες να έρθουν στην αίθουσα. Θα γίνει μια μικρή ανακατάταξη και κατόπιν θα ξαναρχίσουμε μετά από λίγα λεπτά με την ακρόαση. Υπότιτλοι Authorwave Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ώρες μόνο και το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω τους συναδέλφους, τους εμπειρογνώμονες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα τις πολιτικές ομάδες οι οποίες βοήθησαν δημιουργώντας μία ομάδα με μέλη όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Η κυρία Κομίνα απούσα, διότι είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις για το ΕΛΚ, με το ΕΛΚ. Οι συντονιστές λοιπόν δημιούργησαν αυτήν την ε, ομάδα η οποία έχει σαν αποστολή να συντονίσει τις εργασίες εν ώψη της θέσης ισχύ της οδηγίας για το 2005. Μια σημαντική οδηγία για θέματα εξαιρετικά σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ελευθερία υπηρεσιών, αλλά και για το μέλλον της ε, ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Πρόκειται λοιπόν για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και η σημερινή μας ακρόαση είναι ενδεχομένω ένα πρώτο βήμα για τις προτάσεις που θα πρέπει να υποβάλουμε. Θα πρέπει καταρχήν λοιπόν να ξεκαθαριστούν οι κανόνες, να απλοποιηθούν οι κανόνες έτσι ώστε να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσφατη μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία δημοσιεύτηκε και παρουσιάστηκε στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο, υπογραμμίζει και δείχνει ότι όχι μόνο υπάρχει πάρα πολύ σημαντική καθυστέρηση σε όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη μεταφορά αυτής της οδηγίας, αλλά και πρακτικές δυσκολίες οι οποίες έχουν προκύψει από την εφαρμογή της. Συζητούσα πριν λίγο με μια κύρια η οποία μου εξηγούσε ότι υπάρχουν όχι μόνο διαφορετικές πληροφορίες από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, αλλά πολλές φορές και αντιφατικές και αντικρουόμενες. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να εξετάσουμε το θέμα αυτό, γι' αυτό και καλέσαμε ένα μεγάλο αριθμό εμπειρογνωμόνων. Περιμένουμε λοιπόν από τις παρουσιάσεις τους διευκρινήσεις όσον αφορά θέματα νομοθετικά Δεύτερον, αν υπάρχουν και αν έχουν εντοπιστεί δυσκολίες για την ελεύθερη κυκλοφορία και εάν υπάρχουν νέες δυσκολίες και νέα εμπόδια λόγω και εμπόδια κυρίως που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους ειδικού, όλους τους εμπειρογνώμονες. Σας ζητώ, σας παρακαλώ πολύ να περιοριστείτε στο χρόνο ομιλία σας, που είναι 10 λεπτά και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Η κυρία Λούσια Μέστρ, η οποία είναι συντονίστρια στην Πορτογαλία, θα μας μιλήσει για την Πορτογαλία. Ο κύριος Πολ Φίλιπ, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικού για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μας μιλήσει συγκεκριμένα για το προσωπικό, το επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό, η κυρία Rosemary Μακάλιστερ Σμιθ, είναι επίσης παρούσα, ο κύριος Τζέισον Αρούντα. Από το ίδιο Συμβούλιο Εξωτερικές Σχέσεις, ο κύριος Ντάιρον Σέλ, Επικοινωνία και η κυρία Τένσε Σούμπερ, επίσης από τον ίδιο οργανισμό, ιατρικό οργανισμό, και η κυρία Άννα Χόλαντ, από τον ε, φορέα Fitness to Practice. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλιπ. Ο κύριος Αρνό Μέτσνερ από τον ε, Εθνικό Γερμανικό Σύλλογο ο οποίος θα μας μιλήσει για την εμπειρία του στο θέμα αυτού του, ε, αυτής της οδηγίας, ο κύριος Φίλιπ Βόλτερς, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μηχανικών, ο Μάικελ Ντεμπλάστ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και ο Γιένς Μπορναβολτ, σα ζητώ συγγνώμη γιατί πιστεύω ότι δεν προφέρω σωστά το όνομά σας, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την επαγγελματική κατάρτιση, όπως θα μας μιλήσει για την πιστοποίηση όσον αφορά την κατάρτιση, τη διαβίου κατάρτιση και την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Καταρχήν λοιπόν δίνουμε το λόγο στην κυρία Λούσια Μέστ, συντονίστρια για την Πορτογαλία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής αυτής. για την ιστορική αγορά και την πράσπιση των καταναλωτών. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου στείλατε. Επίσης, ε, να χαιρετήσω τους κύριους βουλευτές και τους συναδέλφους που έκαναν σχόλια για την οδηγία του 2005-36. Η δική μου εμπειρία στον τομέα αυτό είναι 15 15 ε, ετών. Εγώ λοιπόν είμαι ένα άτομο που θα μπορούσε να σας μιλήσει για την εμπειρία της εφαρμογής άλλων οδηγίων, ε, κυρίως του γενικού συστήματος ε, και στο στάδιο αυτό τι σημαίνει η οδηγία αυτή για την Πορτογαλία, σε πορτογαλικό επίπεδο. Και θα ξεκινήσω από το εξή. Στην Πορτογαλία εμείς ε, μεταφέραμε στο σωστό μας δίκαιο αυτή την οδηγία μέσω μίας ε, και μόνης ε, πράξης και ουσιαστικά εκεί καλύπτουμε όλα τα επαγγέλματα και του γενικού συστήματος και της αυτόματης αναγνώρισης. Δηλαδή, η οδηγία συμπεριλαμβάνει 15 οδηγίες 13 του Γενικού Συστήματος ε, και 2 που αφορούν την αυτόματη αναγνώριση και στην Πορτογαλία εμείς συμπεριλαμβάνουμε συμπεριλάβαμε ε, σε μία και μόνη πράξη του, με ημερομηνία Μάρτιο του 2009 όλο αυτό το έργο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εδώ ξεκινά η απλούστευση ε, και εμείς στο νέο δίπλωμα έχουμε ε, ουσιαστικά αναφέρουμε ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές στην Πορτογαλία. Έχουμε 35 αρμόδιες αρχές στην Πορτογαλία, 9 υπουργεία και συνολικά μιλάμε για 35 ρυθμισμένα επαγγέλματα ε, εδώ το επάγγελμα ε, των ε, γιατρών στην αυτόματη αναγνώριση σας περιλαμβάνεται όμως εδώ έχουμε μία απλούστευση με αυτό το πλαίσιο γιατί, γιατί και οι πολίτες αλλά και οι αρμόδιες αρχές ουσιαστικά εκεί είδαν ποιες είναι οι διαδικασίες και ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα ποιες είναι οι προθεσμίες όλα αναφέρονται στο ίδιο δίπλωμα και επίσης είναι και πιο απλή η διάρθρωση μεταξύ αρμοδίων αρχών που προηγουμένως δεν γνωρίζονταν, γιατί σε ό,τι φορά την αυτόματη αναγνώριση υπήρχαν επιτροπές. Εκεί συζητούνταν ε, το θέμα της αναγνώρισης αυτών των επαγγελμάτων. Και στην περίπτωση των ε, επαγγελμάτων του Γενικού Συστήματος ε, συζητείται το θέμα εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, έτσι λοιπόν εδώ έχουμε την εφαρμογή και της δεύτερης και της τρίτης οδηγίας η οποία έρχεται να απλουστεύσει όλες αυτές τις οδηγίες καθώς τις ενοποιεί. Λοιπόν, αυτές, αυτή η ανταλλαγή ε, των ε, βαλίτων πρακτιών γίνεται γιατί όταν αρχίσαμε να μιλάμε για μηδέν γνώριση πρέπει να σκεφτούμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει ε, και οι ίδιε οι αρμόδιε αρχέ, στην περίπτωση Πορτογαλία, είναι ουσιαστικά οι ενώσει, οι σύλλογοι των γιατρών, των φαρμακοποιών κτλ. Επίση θα πρέπει να εφαρμόσουν κάποιε διαδικασίε στα πλαίσια του γενικού συστήματο. Θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα αποζημίωση χάρη και έτσι λοιπόν ε, όταν ε, Ινδίας έρχονται σε επαφή με τους ομολόγους τους στο πλαίσιο του γενικού συστήματος, ε, τότε ε, υλοποιείται καλύτερη εργασία. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει ε, ανταλλαγή βέλτιση στον πρακτικών μεταξύ των ε, αρχών, των αρμοδίων αρχών και μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί μεταξύ των κρατών μελών, ε, γιατί ε, η Γενική Διεύθυνση της Ιστορικής Αγοράς δημιουργήθηκε μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που την αποκαλούμε OMI Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία εφαρμόζεται σε ε, όλα ένα και περισσότερα επαγγέλματα και αυτό διευκολύνει πάρα πολύ την αναγνώριση των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών προσόντων Δηλαδή, ε, μία πορτογαλική αρχή, αν έχει αμφιβολίες ε, σε σχέση με μια άλλη αρμοδία άλλου κράτους μέλους, με αυτόν τον εύκολο τρόπο μπορεί μέσω της πλατφόρμας να υπέρβει τα εμπόδια τα οποία, είχα, οποία υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί δεν ήταν γνωστή η άλλη πραγματικότητα. Εγώ, ε, λοιπόν, εδώ αναφέρθηκα στη διαφάνεια, ε, στον επιμερισμό των πρακτικών και μεταξύ κρατών μελών, ε, την εφαρμογή των σημείων επαφής εγώ νομίζω ότι αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εδώ εμείς ε, στην Πορτογαλία ε, χρησιμοποιούμε και την πορτογαλική και την αγγλική γλώσσα για να δημοσιοποιήσουμε όλα τα σημαντικά έγγραφα αλλά και τον κώδικα δεοντολογίας που χρησιμοποιείται μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Ε, υπήρξε ουσιαστικά μελέτη του θέματος αυτού στην ομάδα των συντονιστών. Και μάλιστα αυτό μας επιτρέπει να εντοπίσουμε και μια σειρά βέλτιστων επιθυμητών και αποδεκτών πρακτικών και βέβαια μιλάμε και για ορισμένε απαράδεκτες πρακτικές, ε, για ορισμένα κρατημέλη. Και Παραδείγματο χάρη, μπορεί κάποιο να προσφύγει σε ένα δίκτυο Solvit για να παρουσιάσει μια υπόθεση και στη συνέχεια μπορεί να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ουσιαστικά εδώ φύγω έξι ε, ε, σημεία ε, σχέση με τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Αυτό το μεγάλο στίχημα δηλαδή στον κώδικα διοντολογία αλλά ε, και την εργασία που έγινε για τον εντοπισμό σημαντικών εγγράφων έτσι ώστε ο καθένα να γνωρίζει ε, όταν παραδείγματος χάρη μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος ποια είναι τα σημαντικά έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του και που επιτρέπει ουσιαστικά να μεταφράσει ουσιαστικά τα προσόντα του, γιατί σε κάθε κράτο μόνο υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητε. Και μέσω από αυτή την ταυτοποίηση είναι πιο εύκολο ο πολίτης να εντοπίσει συγκεκριμένα προβλήματα ή τουλάχιστον να επιλύσει πολλά από τα προβλήματά του. Ε, έχουμε επίσης και τον οδηγό του χρήστη που θα είναι σύντομα στην ιστοσελίδα. και έχουμε ουσιαστικά ένα σύνολο ερωτήσεων και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Αυτό ο οδηγός θα είναι πάρα πολύ σημαντικός όχι μόνο για την αρμόδια αλλά και για τον ε, ίδιο τον πολίτη, το μετακινούμενο. Τώρα, σε σχέση με την στήριξη στη συνιστόσα της παροχής υπηρεσιών, αυτή είναι μία συνιστόσα καινοτόμο στο σύστημα της αναγνώρισης. Λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη της οδηγίας των υπηρεσιών και επίσης θέλουμε να διευρύνουμε και το σύστημα είμαι στο ε, και στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Ο χρόνο είναι πάρα πολύ λίγο, αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω και μια σειρά προτάσεων που νομίζω ότι μπορούν να είναι αυτές ε, που θα μπορέσουν να απασχολήσουν κάποια κράτη-μέλη. Αλλά μπορεί ορισμένε από αυτέ τι ε, προτάσει και υποδείξει να σα βοηθήσουν να επιλύσετε κάποια αναπομείναντα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι ένα τμήμα τη διάδοση, τη δημοσιοποίηση αυτών των θεμάτων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ε, είναι ε, πολύ σημαντικό στο δίκτυο Solvit και EURES. Ε, εγώ προσωπικά βλέπω ότι στο πόρταλ, στην πύλη του δικτύου EURES δεν ε, αναφέρονται με σοφήνεια, τα σημεία επαφής, ε, δηλαδή παραδείγματο χάρη δημοσίευεται μία προσφορά εργασίας, αλλά ε, ουσιαστικά ο πολίτης δεν ε, καταλαβαίνει πού πρέπει να παρουσιάσει την αίτησή του, ούτε κατανοεί ότι υπάρχουν προθεσμίες που μπορεί να τρέχουν για τρει τεσσερις μήνες και μάλιστα μπορεί να εφαρμόζεται και ένα μέτρο, παραδείγματο χάρη, όπω το να περάσει από μια πρακτική, από ένα στάζ. εγώ νομίζω ότι είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και τα δύο και το Solvit και το να δίνουν ε, ουσιαστικά δημοσιοποίηση, να δημοσιεύουν όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν αυτή την οδηγία και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Τώρα, συνέχεια το να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία πλατφόρμων και αυτό είναι ένα μέσο να υπερβληθούν τα εμπόδια. Υπάρχουν ε, ουσιαστικά κάποια εμπόδια που συνίσταται στην ύπαρξη μέτρων αποζημίωσης. Ε, ουσιαστικά μπορεί να μπλοκάρουν την αγορά. Έτσι λοιπόν πρέπει να δώσουμε κίνητρα για τη δημιουργία αυτών των κοινών πλατφόρμων. Πρέπει να εφαρμοστεί ένα δίκτυο σημείων επαφής που να είναι αποτελεσματικό και πρέπει να υπάρχουν τακτικές συνεδριάσεις, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, Παραδείγματο χάρη μπορεί να υπάρχουν συνεδριάσει και κατά τη διάρκεια ε, των προεδριών. Ε, στη σημερινή, στη μελλοντική προεδρία, παραδείγματο χάρη, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα σημεία επαφή να καλέσουν τις αρμόδιες αρχές και να ανταλλάξουν ε, τις αμφιβολίες τους και τους δασμούς τους στο επίπεδο αυτό. Γιατί, εντάξει, έχουμε αφενός τις συναντήσει στι Βρυξέλλε, όμως αυτό είναι το ένα και είναι διαφορετικό τα σημεία επαφή να ε, μεταβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες στη χώρα τους. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διάρθρωση μεταξύ αυτής της οδηγίας και της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Εγώ νομίζω ότι εδώ ε, πρέπει να γίνουν σεμινάρια, εκδηλώσεις, ε, κοινέ και θα περάσω στο σημείο 5 και 6. Πέμπτον, συντονισμό τη οδηγία πρέπει να μα επιτρέψει συνεχή επικαιροποίηση τη βάση δεδομένων. Αν ε, εγώ είχα υπαρκή χρόνο, θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε ε, ποιος έχει βάση δεδομένων και θα γνωρίζαμε ποια είναι τα ρυθμισμένα επαγγέλματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα γνωρίζαμε ε, σε κάθε ένα από τα, για κάθε ένα από αυτά τα επαγγέλματα ποια είναι η αρμόδια αρχή στην οποία πρέπει να απευθυνθεί ο πολίτη. Και τέλο, θα μπορούσαμε να γνωστοποιήσουμε τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ τη οδηγία τη ακαδημαϊκή αναγνώριση και του ευρωπαϊκού πλαισίου αναγνώριση των προσόντων. Γιατί γνωρίζουμε ότι έχουν ανακύψει προβλήματα εκεί. Έτσι λοιπόν αυτές οι ε, τελευταίες συστάσεις ε, θα πρέπει ε, να υλοποιηθούν προκειμένου να απλουστευτεί η οδηγία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μπόρεσα να συνεισφέρω με κάποιες προτάσεις που θα μπορούσατε να τις λάβετε υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας. Θα δώσω μέσα στο λόγο τον Πολ Φίλιπ, του ε, Γενικού Συμβουλίου του Ιατρικού των, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτό το θέμα. Λέγομαι Πολ Φίλιπ, εκπροσωπώ το Γενικό Ιατρικό ε, Συμβούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η ρυθμιστική αρχή και τα θέματα που μας αφορούν είναι θέματα ασφάλειας για τους ασθενείς. Ε, δεν ε, έχουμε, αν θέλετε, εκπροσώπηση άλλου είδους των ιατρών στη χώρα μας, αλλά κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια και η προστασία των ε, ασθενών. Επίσης, διατηρούμε ένα μητρό των ε, ατόμων που ασκούν το επάγγελμα του γιατρού στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει κάποιων ε, προτύπων και σκοπός αυτού του Μητρώου είναι τα μέλη μας να διασφαλίζουν ε, την ε, προστασία και την ασφάλεια των ασθενών. Υπάρχουν 230.000 ε, γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στα μητρώα μας και οι οποίοι εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην χώρα μας, όπως ξέρετε, μάλλον εισάγουμε παρά εξάγουμε γιατρούς. Εργαζόμαστε σε συνεργασία, σε εταιρική σχέση με άλλες ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ομάδες και φορείς που επίσης, όπως και εμείς, εργάζονται με σκοπό την προστασία του κοινού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συνεργασία είναι σε θελοντική βάση, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητική και ότι βεβαίως υπάρχει ε, μια καλύτερη κατάσταση σήμερα. Μας απασχολούν θέματα όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, ιατρών αλλά και των ασθενών. Επαναλαμβάνω ότι στο επίκεντρο της προσοχής μας βρίσκεται η ασφάλεια και η προστασία των ασθενών, αλλά προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τις δυνατότητες κυκλοφορίας των ασθενών, εάν, εάν βεβαίως υπάρχουν εγγύησεις για την προστασία και την ασφάλειά τους. Εδώ υπάρχει βεβαίως μια αντιφατική θα έλεγα τάση μεταξύ της υψηλής προστασίας της παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας υψηλής ποιότητας, της ασφάλειας δηλαδή και της προστασίας των ασθενών και της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών από το ένα κράτος στο άλλο. Και η οδηγία η οποία συζητείται σήμερα σαφώς και ε, μπορεί σε κάποια σημεία να επιδεινώσει την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών. Οι προκλήσεις είναι πολύ σημαντικές Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, χρειάζεται εμπιστοσύνη, αμοιβαία κατανόηση ότι υπάρχουν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, παραδείγματο χάρη. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιαίτερα σε διάφορους τομείς επαγγελματικούς, όπου είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο η διασυνοριακή συνεργασία, αλλά και η κυκλοφορία των ασθενών. Χρειάζεται λοιπόν ρύθμιση, χρειάζεται διαφάνεια, πρέπει να υπάρχουν μητρώα για τους ιατρούς, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο και από άλλες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών, έτσι ώστε να υπάρξει, όπως σας είπα, διαφάνεια και την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει σε μία τακτική βάση να μπορούν να ε, ανταλλάξουν πληροφορίες, ενημέρωση και να υπάρχει και δυνατότητα προσφύγης ε, στα δικαστήρια εάν υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις ε, των κανόνων και των ρυθμίσεων η υποχρέωση για παραδείγματο χάρη ανταλλαγή πληροφοριών εάν υπάρχει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας ή για εσφαλμένες πρακτικές, εάν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών, Εμείς έχουμε δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών. Πιστεύω ότι μέσω των πρωτοβουλειών για τη διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων να βελτιωθεί. Και πιστεύω ότι στις 2 Δεκεμβρίου θα πρέπει να συζητηθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το σύστημα που υπάρχει, το IMIS, το οποίο βεβαίως και μπορεί να βελτιωθεί αλλά πιστεύω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει με ευελιξία να υποβληθούν σε αυτήν την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει μέσω αυτής της ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών οι αρμόδιες αρχές να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και δεσμευτικό σύστημα και ζητάμε εδώ να ενημερωθεί το σύστημα, να υπάρξει ένα μητρό το οποίο να βασίζεται όχι μόνο στα σφάλματα και στις παραβιάσεις που έχουν ε, εξεταστεί, αλλά στις αρμοδιότητες, στα προσόντα και να υπάρχει και ένα σύστημα ασφαλιστικό όσον αφορά την πιστοποίηση αυτών των αρμοδιοτήτων και προσόντων. Τελειώνοντας, πιστεύω ότι θα πρέπει σε πολλά σημεία να αναθεωρηθεί το κείμενο της οδηγίας. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει καμία διάταξη που να επιτρέπει τον οποιοδήποτε έλεγχο σε έναν γιατρό, σε έναν επαγγελματία, πριν του δοθεί η άδεια να εγγραφεί στα Μητρώα. Υπάρχει μία πρόβλεψη, η οποία όμως κατά την άποψή μας δεν αρκεί και είναι και ασαφής. Αυτά ήθελα να σας πω σαν εισαγωγικά σχόλια, αλλά βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας εάν θέλετε να ε, κάνετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Eh Κύριε Μα είπατε πάρα πολλά σε 7 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν επιτρέψατε όχι στον επόμενο να ε, μακρηγορήσει για 12 λεπτά, αλλά ίσως θα επιτρέψει στη συζήτησή μας να είναι πιο πλούσια γιατί θα έχουν την ευκαιρία περισσότερο να μιλήσουν. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την παρέμβασή σα Και φυσικά μην ε, φοβάστε, σίγουρα θα απευθυνθούμε σε ο κύριος Μετσέ τώρα από την Γερμανική, Γερμανική, Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση θα μας δώσετε πληροφορίες για την εμπειρία των μελών, για την εφαρμογή της οδηγίας στη Γερμανία, γιατί ουσιαστικά εκπροσωπείτε ε, τους ελεύθερους Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην Δανία, ε, στη Γερμανία έχουμε ε, ένα ε, ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες ε, και εκπροσωπώ την ε, ένωσή τους ε, και μιλάμε για ρυθμισμένα και μη ρυθμισμένα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι, τα περιφερειακά επιμελητήρια που είναι αρμόδια και για τα ρυθμισμένα επαγγέλματα εξετάζουν δηλαδή τα επαγγελματικά προσόντα των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζουν δηλαδή τα προσόντα και την ποιότητα της δουλειάς των ε, επαγγελματιών. Ο ασθενής, ε, για παράδειγμα, δεν είναι σε θέση να εξετάσει την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει. Το ίδιο ισχύει για ε, τον πελάτη ενός αρχιτέκτονα, για παράδειγμα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να συμμετέχουμε, να συμμετέχουμε ε, στο Solvit και υπάρχουν πολλά ερωτήματα στον τομέα αυτών. Ήθελα όμως να πω ανοιχτά επίσης ότι λίγα προβλήματα έχουμε τα οποία δεν μπορούμε να λύσουμε. με την οδηγία αυτήν ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε ε, είναι οργανωμένοι σε περιφερειακό επίπεδο. και ε, γενικά οι επαγγελματίε μα κινούνται σε, ένα, σε ακτίνα 25 μέχρι 200, μέχρι 200 χιλιόμετρα. Ε, υπάρχουν ε, δηλαδή κάποιε περιπτώσει που ξεπερνούν τα σύνορα ενό κρατηδίου. Υπάρχει το θέμα των ασφαλίσεων, υπάρχει το, των επαγγελματικών ασφαλίσεων, υπάρχει το θέμα της γλώσσας και της κουλτούρας. Όλα αυτά δεν είναι ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό είναι δύσκολο να παρέχει κανείς υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, κάποιος επαγγελματίας που έρχεται στη Γερμανία δεν είναι πολύ εύκολο ε, να συμμετέχει στο ε, ε, εθνικό σύστημα υγείας. Το ίδιο ισχύει και για Γερμανούς γιατρούς που πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Εκπροσωπούμε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι ο ελεύθερος επαγγελματία ενεργεί σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο σημαίνει ε, θα πρέπει να γνωρίζει ξένες γλώσσες κλπ. Και φυσικά θα πρέπει να γνωρίζει τις αγορές στις ε, οποίες θέλει να δραστηριοποιηθεί, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ε, ανθρώπων στους οποίους θέλει να παρέχει τις υπηρεσίες του. Οι δικηγόροι και οι λογιστές ε, δεν, ε, ε, δεν ενεργούν τόσο πολύ διασυνοριακά όσο για παράδειγμα οι όσο οι αρχιτέκτονες. Και υπάρχουν διάφοροι επαγγελματίε οι οποίοι θα πρέπει να ε, κάνουν κάποιε εξετάσει για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν σε άλλη χώρα. Στην ε, Γερμανία. Λοιπόν, ε, βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες κυρίως επαγγελματιών δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. Η οδηγία ε, αυτή, αυτή ε, από πλευρά δομή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο. Διαπιστώνουμε όμως επίσης ότι η εφαρμογή δεν γίνεται πάντα με άψογο τρόπο, για να το πω ευγενικά κιόλα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν καλύτερα να συντονιστούν καλύτερα και μπορούν με οδηγίες ή με διαφορετικές διατυπώσεις να βελτιώσουμε την εφαρμογή της οδηγίας. Συμπέρασμα, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ψάχνουμε για μια προσέγγιση και επιδιώκουμε τη βελτίωση της εφαρμογής οδηγία. οδηγίας. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω εδώ τρία βασικά στοιχεία. Καταρχήν, σημαντικό για μας είναι να συζητιέται το θέμα της εκπαίδευσης. Ε, μπορώ να αναφέρω τη διαδικασία της Πολόνια. Διαπιστώνουμε επανειλημμένα ότι κάποιος που ε, είναι μηχανικός ε, δικηγόρος, αρχιτέκτονας ε, στην Γερμανία και ψάχνει κάποιον συνεργάτη, δεν ψάχνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός λοιπόν να μπορεί να αξιολογήσει σωστά τα προσόντα κάποιου άλλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, εξετάζουμε την ποιότητα και να βελτιώσουμε τις ε, διασυνοριακές υπηρεσίες. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, να μην έχουμε διαφορετικά πρότυπα. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο επίπεδο ποιότητας και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ανταγωνισμό στην ποιότητα προς τα πάνω, να επιδιώξουμε βελτίωση της ποιότητας. Επίσης, είναι σημαντικό να είναι όλα αυτά γνωστά στο κοινό. Ήδη ανέφερα ότι είμαστε σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές και οι διευθυντές προσωπικού θα πρέπει να γνωρίζουν βέβαια πώς θα αξιολογήσουν τα προσόντα κάποιου άλλου. Θέλουμε όμως και οι καταναλωτές να γνωρίζουν πώς έχει η κατάσταση. Στη Γερμανία κάναμε έρευνες σχετικά με το τι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές στην παροχή υπηρεσιών. Και ε, το 96% είπαν ότι, ε, θέλουν, ε, ε, ότι είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα, με τα προσόντα. Δεν θέλουμε λοιπόν να επιδρώσουμε την κατάσταση, θέλουμε να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό. Η αξιολόγηση των ανθρώπων γίνεται με επαγγελματική και όχι με προσωπικά κριτήρια. Για παράδειγμα, δεν τίθεται θέμα ποινικού μητρώου. Για μας αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Διότι θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη των ε, πελατών προς το πάροχο των υπηρεσιών. Επίσης ε, θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο το θέμα του κώδικα της δεοντολογίας και θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να, να ε, συμπεριλάβουμε εδώ και το θέμα της προστασίας των δεδομένων και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα παλιό αίτημα της Ένωσής μου να υπάρχει ένα κεντρικό μητρό για παραβάσεις. Δεν θα συμπεριλαμβάνει βέβαια κάτι τέτοιο όλα τα επαγγέλματα, ε, αλλά τουλάχιστον τα ρυθμισμένα. Οι εμπειρίες που έχουμε κάνει και φτάνω στο τέλος της παρέμβασής μου, το συμπέρασμα είναι ότι η οδηγία αυτή επιφέρει σαφώς θέμενη αξία. Είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή κοινότητα το θέμα αυτό. Το θέμα είναι πόσο βελτιώ... μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να λύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Πιστεύω ότι η οδηγία αυτή θα αποτελέσει θετικό στοιχείο και δεδομένων των ε, προβλημάτων που υπάρχουν. Ε, πιστεύω ότι σε δύο-τρία χρόνια θα πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία αυτή με βάση τις ε, εμπειρίες που θα έχουμε συλλέξει στο μεταξύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φιλίπ Πότερς, ε, που είναι Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Συλλόγων Μηχανικών και θα μας σχολιάσει τις εμπειρίες των μηχανικών στα διάφορα κρατημέλη σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργεί η αμοιβή αναγνώριση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που καλέσατε τη ΦΕΑΝΗ, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Συλλόγων Θα ήθελα η παρουσίασή μου τη δούμε, να σας πω ότι εγώ εργάζομαι στην βιομηχανία, είμαι πτυχούς μηχανικός και εδώ και 10 χρόνια είμαι γενικός γραμματέας αυτής της ομοσπονδίας, όπως ε, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στις ε, διαφάνειες που θα τις παρουσιάσω. Ε, θα είναι στα αγγλικά, γι' αυτό και εγώ θα μιλήσω αγγλικά. Λοιπόν, Μάλλον ε, να πω δύο λόγια για τη Φεάνη, έτσι ώστε να γνωρίζουν ε, όλοι περί τίνος πρόκειται και στη συνέχεια θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες ε, για την κατάρτιση των μηχανικών και για το πώς ρυθμίσετε το επάγγελμα και τους διάφορους μηχανισμούς που υπάρχουν για τη βελτίωση της αναγνώρισης και στη συνέχεια για να φτάσουμε στο συμπέρασμα. Φέανη λοιπόν είναι μια ομοσπονδία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 να συνεχίσω στα γαλλικά μάλλον αφού το ξεκίνησα. Η ΦΕΑΝΗ ουσιαστικά συγκεντρώνει όλες τις ε, εθνικές ε, νόσεις μηχανικώ. Ε, τώρα είμαστε 30 χώρες και η Ρωσία συμμετέχει. Ουσιαστικά συμμετέχουν 350 εθνικές οργανώσεις και 3,5 εκατομμύρια μηχανικοί στόχοι της ΦΕΑΝΗ πάντοτε ήταν η βελτίωση της κινητικότητας, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και στο πλαίσιο αυτό η οδηγία μας ε, διευκολύνει φυσικά σε αυτή τη δραστηριότητα. Κάναμε λοιπόν μία μελέτη για ε, το, εγκατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ βλέπετε τις πληροφορίες που αναλύθηκαν και ε, δεν υπάρχουν δύο χώρες στην Ευρώπη που να έχουν το ίδιο σύστημα για τους μηχανικούς και που να έχουν την ίδια διάρκεια ως προς την κατάρτιση, την εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, αν συγκρίνουμε ε, τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφορών χωρών, ε, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση και βλέπετε εδώ τα διπλώματα και τους τίτλους ε, που δίνονται από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαφέρουν ε, οι τίτλοι, έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να τα συγκρίνουμε όλα αυτά. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πρέπει λοιπόν ε, να βλέπουμε ότι έχουμε δύο είδη μηχανικούς. Έχουμε τον μικρό, το σύντομο κύκλο και το μεγάλο κύκλο. Ε, τώρα, σύμφωνα με την ορολογία της Μπολόνια, έχουμε τον bachelor και το master. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι στην Ευρώπη ο πρώτος κύκλος δεν αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες. Δηλαδή, τα άτομα που έχουν ε, κάνει τις σπουδές αυτές δεν μπορούν να ασκήσουν ε, το επαγγελμα του μηχανικού. Επίσης αναλύσαμε το πώς ρυθμίζεται το επάγγελμα στην Ευρώπη και όπως βλέπετε στο βορρά ε, με το λευκό δεν είναι καθόλου ρυθμισμένο το επάγγελμα, δηλαδή μπορεί κάποιος να σκεφτεί το επάγγελμα χωρίς να έχει λάβει κατάρτιση, όμως ε, στις ε, χώρες του Νότου έχουμε πολύ μεγάλη ρύθμιση, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να το σκέσει χωρίς να έχει την άδεια των εθνικών αρχών, περνά δηλαδή εξετάσεις και πρέπει να γραφεί στο σύλλογο και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης η ρύθμιση εξαρτάται από το τι δουλειά ακριβώς κάνει ο μηχανικός. Επίσης, ενδιαφέρον να ξέρουμε είναι τα στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν 4 εκατομμύρια επαγγελματίες στην Ευρώπη. Έχουμε εδώ πηγές από την Ευρωστάτ και το 85% απασχολείται σε επιχειρήσεις και μόνο το 15% είναι αυτοαπασχολούμενοι ή ε, πάροχοι υπηρεσιών, όπως βλέπετε εδώ. Όταν ε, αναλύουμε την κινητικότητα των μηχανικών, ε, είναι πολύ μικρή, πολύ λίγη ουσιαστικά δεν είναι Μιλάμε περίπου για 500.000 το χρόνο. Λοιπόν, αν τα δούμε όλα αυτά, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, βλέπουμε ότι Έχουμε μεγάλη κινητικότητα στους ε, ε, υπαλλήλου ε, και πολύ λίγη κινητικότητα στους αυτοαπασχολούμενους. Και στο κεντρικό τμήμα που βλέπετε ρυθμισμένα επαγγέλματα, ρυθμισμένο επάγγελμα, υπάρχει μικρή κινητικότητα και βλέπουμε ότι μιλάμε περίπου για 1.750 μηχανικούς που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία ετησίως. Επίσης, όπως είπαμε και προελίσσετε, πρέπει να δούμε το εξή ότι η αναγνώριση των προσόντων σήμερα βασίζεται στην ε, ποσότητα των μαθηματικών, της φυσικής, των μαθημάτων που έχει δηλαδή λάβει κανείς και δεν βασίζεται στις ε, ικανότητες που έχει αποκτήσει, αλλά στο πώς αποκτήθηκαν αυτές οι ικανότητες. Εδώ βλέπετε πώς γίνεται η αναγνώριση των προσόντων. Έχουμε ε, το 60% των μηχανικών ε, που έχουν σπουδάσει 6 χρόνια και οι περισσότεροι αναγνωρίστηκαν, ε, το 4% μετά από ένα τεστ και περίπου 23% μετά από κατάρτιση. Δηλαδή το 90% των μηχανικών αναγνωρίζονται από το ένα σύστημα στο άλλο. Και τα αρνητικά είναι τα εξή. Έχουμε 11%. Δηλαδή, η συνάρνηση δηλαδή Μπορούμε λοιπόν να θέσουμε την εξή ερώτηση. Υπάρχει πράγματι σοβαρό πρόβλημα αναγνώρισης των προσόντων μηχανικών στην Ευρώπη. Είναι κάπως ε, αρκετά περιθωριοποιημένο. Και επίσης ε, η ερώτηση είναι αν η οδηγία βελτιώνει σήμερα και στο μέλλον αυτή την αναγνώριση των προσόντων. Η οδηγία προσφέρει ε, κάποια εργαλεία για τη βελτίωση της αναγνώρισης. Ε, έχουμε καταρχήν το τμήμα του την κοινή πλατφόρμα και την επαγγελματική κάρτα. Θα δούμε ε, αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε το τμήμα και το παράρτημα καθώς υπάρχουν διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα είναι πρακτικά αδύνατο να συμφωνηθεί ένα τμήμα και ένα παράρτημα και ε, να συμφωνηθεί ο κατάλογος των μαθημάτων. Έτσι, λοιπόν, θα έπρεπε αυτό το τμήμα και το παράρτημα να γίνει αποδεκτό σε όλους και αυτό ξεχάστε το. Έτσι λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα για την κοινή πλατφόρμα. Εδώ μελετήσαμε λεπτομερώς τη δυνατότητα αυτή. Εδώ να πούμε ότι αυτή η κοινή πλατφόρμα θα έπρεπε να δημιουργήσει κάποιες γέφυρες. Ε, όμως, στην περίπτωση των μηχανικών δεν μιλάμε για ένα επάγγελμα. Υπάρχουν ε, πολλαπλά είδη κατάρτισης. Έτσι λοιπόν, πώς θα έχουμε μια πλατφόρμα για ένα συγκεκριμένο ε, επάγγελμα. Αυτό μας εμποδίζει να περάσουμε από το ένα επάγγελμα στο άλλο και τελικά μάλλον θα μειωθεί η κινητικότητα παρά θα αυξηθεί. Επίσης, ε, όπως αναλύσαμε, είναι πρακτικά αδύνατο τεχνικά να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα για τους μηχανικούς. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κινούμενο στόχο και δεδομένης προσπάθειας που θα πρέπει να γίνει ε, και λαμβάνοντας υπόψη το ότι δεν έχουν πολυμηχανική πρόβλημα, τελικά ε, απορρίψαμε και αυτή την επιλογή. Επομένως, μένει η επαγγελματική κάρτα. Και εδώ να σας αναφέρω, ε, σας αναφέρω εδώ ένα κείμενο της οδηγίας λέγεται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διευκολύνει την ε, αναγνώριση αν ε, υπάρχει ουσιαστικά μια ε, σειρά ουσιαστικά δεδομένων. Εδώ βλέπετε το επαγγελματικό πλαίσιο στα δεξιά με το νέο. Αυτό το νέο έχει ενταχθεί σε αυτό που έχει προτείνει η Κομισιόν για την κάρτα Europass. Όλα λοιπόν είναι εφικτά. Έχουμε κάνει και μια μελέτη σκοπιμότητας. Μελετήσαμε όλα τα είδη της κινητικότητας ε, και ε, τα αιτήματα και των μηχανικών και των εθνικών δικήσεων και των ε, εργοδοτών. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρώτον είναι αδύνατο να εκτιμήσουμε το πόσο θα βελτιωνόταν η κινητικότητα των μηχανικών, γιατί δεν γνωρίζουμε ε, γιατί αν έχουμε 10% δεν έχουμε παραπάνω, δηλαδή γιατί φοβούνται, ε, γιατί δεν θέλουν να φύγουν, φοβούνται ότι δεν πρόκειται να αναγνωριστούν τα προσόντα τους, δεν γνωρίζουμε. Όμως εκτιμούμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση στη γεννητικότητα. Όμως θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια κάρτα επαγγελματική για τους μηχανικούς, όχι μόνο χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Και αυτό θα ήταν ε, ουσιαστικά σαν ε, ένα κατατεθέν ποιότητα για τους Ευρωπαίους μηχανικούς και αυτό θα διευκόλυνε την πρόσληψη των νέων μηχανικών και φυσικά πρόκειται και για ένα μέσο διαφάνειας, ένα εργαλείο διαφάνειας. Σημερασματικά λοιπόν να πω ότι θα θέλαμε η Κομισιόν να συνεχίσει ουσιαστικά τις προσπάθειες που καταβάλει για τη δημιουργία αυτής της επαγγελματικής κάρτας. Ε, υπάρχει ε, ουσιαστικά ένα περιορισμένο αριθμό χωρών όπου πρέπει να σταθεί. Πρέπει να έχουμε πολιτική υποστήριξη Κομισιόν, έτσι ώστε να έχει βάρος αυτή η κάρτα και να αναγνωρίζεται όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωση και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για την οδηγία για τους μηχανικού, περισσότερο αποτελεί ένα quo σε σχέση με το παρελθόν. Επίση, ε, σήμερα νομίζω ότι ουσιαστικά εκφράζει εδώ περισσότερο τη ε, θέση των χωρών που ρυθμίζουν το επάγγελμα και αυτή η οδηγία για τους μηχανικούς ε, ουσιαστικά δεν βελτιώνει σημαντικά την αναγνώριση των προσόντων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτήν την πολύ λεπτομερή παρουσίαση. Κάνατε μια έκκληση ζητώντας την πολιτική στήριξη. Ξέρετε ότι εδώ στην Επιτροπή τη δική μας έχετε βουλευτές που είναι παρόντες οι οποίοι θα σας στηρίξουν. Θα σας βοηθήσουν ψήμ, θα υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο θα βοηθήσει. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Μισελ Ντεμπρούστ, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω στα αγγλικά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε τη δυνατότητα στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά γενικότερα στον τομέα του τουρισμού, να σας κάνουν μια σύντομη παρουσία σήμερα το ε, απόγευμα εδώ. Εκπροσωπούμε κυρίως πράκτορες σε εθνικό επίπεδο, 27 δηλαδή συλλόγους, ενώσους, ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποψήφιες χώρες, όπως από την Κροατία, Ελβετία και Νορβηγία. Ο κλάδος μας κυρίως αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 80.000 επιχειρήσεις, μέλη. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες ε, πολυεθνικές, όλοι τις γνωρίζετε. Thomas Cook, Carlson, American Express, ETUI. Δεν ε, κάνω διαφήμιση αυτών των επιχειρήσεων, απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια ονόματα που σίγουρα όλοι γνωρίζετε. Μεγάλες όμως επιχειρήσεις είναι πολύ λίγες στον κλάδο μας, οι περισσότερες είναι μικρομεσαίες και συνήθως είμαστε παρόντες σε ένα ή δύο μόνο κράτη-μέλη. Οι υπάλληλοι μας φτάνουν το μισό εκατομμύριο και όσον αφορά τον κύκλο εργασιών μας για το 2008, μιλάμε για 310 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα επαγγελματικά προσόντα, ο προηγούμενος ομιλητής που κάθεται και δίπλα μου παρουσίασε τους μηχανικούς. Και αν είχαμε παρουσιάσει γεωγραφικούς χάρτες, νομίζω ότι θα είχαμε παρουσιάσει τους ίδιους. Πρόκειται για μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ρύθμιση τους εξαρτάται από το νομικό σύστημα και από την παράδοση των κρατών μελών. Υπάρχουν χώρες όπως η Ρουμανία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ελλάδα, η Αυστρία, όπου υπάρχει ρύθμιση. Χρειάζεται άδεια, χρειάζονται επαγγελματικά προσόντα για να υπάρξει πρόσβαση στο επάγγελμα του ταξιδιωτικού πράκτορα. Στη Γερμανία, τη Φιλανδία, τις σκανδιναβικές χώρες, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν χρειάζεται να έχουν ειδικέ επαγγελματικές ικανότητες και προσόντα και παρόλη την μεταφορά της οδηγίας η αλλαγή ήταν ελάχιστη όσον αφορά την ομοθεσία. Κυρία Γκέπχαρτ, η οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες ουσιαστικά επηρέασε περισσότερο τον κλάδο μας παρότι η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι η ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι tour operators δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά σημαντικά προβλήματα από τη στιγμή που ε, η οδηγία αυτή μεταφέρεται στα εθνικά συστήματα το 2007. Οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες λειτουργούσαν στα κράτη-μέλη έτσι και αλλιώς είχαν άδεια άσκησης επαγγέλματος, δεν υπήρχαν λοιπόν σημαντικές αλλαγές. Όσον αφορά δε τις μικρές εταιρείες, τις μικρομεσαίες εταιρείες, αυτές συνεχίζουν να ε, εργάζονται σε ένα μόνο κράτο μέλος, άρα δεν έχουν ε, σημαντικές δυσκολίες με τη νέα οδηγία. Όπως ξέρετε, στον δικό μας τομέα η ελεύθερη κυκλοφορία δεν αφορά την επιχείρηση, αφορά τον πελάτη μας. Αυτός ταξιδεύει, αλλά δεν έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή την οδηγία, γιατί όλα πάνε καλά. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ε, στα επόμενα τρία λεπτά θα σας αναφέρω κάποια προβλήματα που υπάρχουν παρόλα αυτά όπως ξέρετε ένας ε, tour operator οργανώνει ταξίδια. Οργανωμένα ταξίδια. Με την συμμετοχή ξεναγών είτε ατόμων που συμμετέχουν και καθοδηγούν αυτά τα οργανωμένα ταξίδια. 180 εκατομμύρια τέτοια οργανωμένα ταξίδια πουλήθηκαν πέρσι σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή πολλών Ευρωπαίων τουριστών γιατί θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα οργανωμένο ε, ταξίδι με άτομα που μιλούν την γλώσσα τους, δεν θέλουν να αφαιθούν στην χώρα την οποία επισκέπτονται με την ε, υπηρεσία και της υπηρεσίες αυτής της χώρας. Συνήθως τα άτομα που ε, ζητούν αυτά τα οργανωμένα ταξίδια είναι ηλικιωμένα άτομα και συχνά αυτά τα οργανωμένα ταξίδια έχουν κάποιο πολιτιστικό περιεχόμενο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τους λεγόμενους ξεναγούς ή managers Και όπως ξέρετε, η οργάνωση αυτού του επαγγέλματος, του ξεναγού, είναι τελείως διαφορετικό από τη μία χώρα στην άλλη. Στην Νότια Ευρώπη είναι πολύ ρυθμισμένο το επάγγελμα, στη Βόρεια Ευρώπη όχι. Στην ε, Ισπανία, στην Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο χρειάζεται άδεια για τους ξεναγούς, όχι για τη Γερμανία, τις σκανδιναβικές χώρες ή την Τσεχία. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε ξεναγούς. Ο λόγος είναι απλός. Η παροχή μιας ε, υπηρεσίας στην γλώσσα που καταλαβαίνει ο συμμετέχουν σε αυτό το οργανωμένο ταξίδι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Στη Ρώμη, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας ε, Λιθουανός ε, ξεναγός είτε στη Μαδρίτη, είτε κάποιος ο οποίος μιλάει τη γλώσσα της Μάλτας στο Παρίσι. Πριν υιοθετηθεί αυτή η οδηγία, η κατάσταση με τους ξεναγούς ήταν περίπλοκη, καθότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζαν τους δικούς τους κανόνες και κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στο νότο της Ευρώπης, επιβάλλεται ο ξεναγός της χώρας, άσχετα με το ποια γλώσσα μιλάει ο ξεναγός αυτός και αν είναι κατανοητή στους συμμετέχοντες στο ταξίδι. Αυτό το 1991 οδήγησε σε μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την οποία τέσσερις χώρες αναγκάστηκαν να αποδεχτούν την απόφαση ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες, ε, τα ίδια προσόντα στον ξεναγό, ο οποίος προσλαμβάνεται επί τόπου με αυτόν τον οποίο μπορεί να προσφέρει το ταξιδιωτικό πρακτορείο. Ιδιαίτερα κοιτώντας κάποιες διατάξεις, αλλά πιο συγκεκριμένα το άρθρο 5 της οδηγίας, βλέπουμε την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος από κάποιον ξεναγό άλλης χώρας σε προσωρινή βάση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την επίσκεψη σε μνημεία τουριστικά είτε μουσεία μιας άλλης χώρας. Και εδώ υπάρχει και μία σημείωση ανεπίσημη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007 που αφορά το θέμα αυτό. Σήμερα η κατάσταση είναι η εξής. Κάποια κράτη-μέλη συνεχίζουν να περιορίζουν την δραστηριότητα ε, αλλοδαπών ξεναγών, οι οποίοι, και θα το πω με διπλωματικό τρόπο, αντιμετωπίζουν ακόμα ε, κάποιες διοικητικές δυσκολίες. Εμείς σήμερα πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτές ε, τις περιπτώσεις της μη αναγνώρισης των προσόντων σε τοπικό επίπεδο. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο ε, εθνικό δίκαιο. Πρόκειται και για την δυσκολία επικοινωνίας και συνεννόησης με τις τοπικές αρχές για τα θέματα αυτά. Οι δυσκολίες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην έλλειψη γνώσης της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην κάθε χώρα. Και πολλές φορές οι εθνικές και τοπικές αρχές δεν γνωρίζουν ε, την νομοθεσία η οποία είναι εφαρμοστέα κάθε φορά. Θα πρέπει λοιπόν εδώ οι εθνικές αρχές να ενημερώσουν τις τοπικές αρχές όσον αφορά την ε, ρύθμιση, την νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα των ξεναγών, ποια είναι τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται, κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει ιδιαίτερα τα 15 εκατομμύρια των Ευρωπαίων που συμμετέχουν σε αυτά τα οργανωμένα ταξίδια κάθε χρόνο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Σα ευχαριστώ και την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι όντω μα δώσατε κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μα οδηγήσουν σε άμεση δράση. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Γιέντ Μπόρνεβολτ. Ζητώ συγγνώμη γιατί προφορά το όνοματά σα. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο του οργανισμού για την επαγγελματική κατάρτιση, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ευρωπαϊκή επιστοποίηση όσον αφορά την εκπαίδευση και την διαβίου κατάρτιση. Σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου ε, Δεξιοτήτων επαγγελματικών προσόντων, που είναι ένα μέσο το οποίο συνδέεται με την οδηγία και νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη σχέση αυτή και να δούμε κατά πόσο τα δύο μέσα αυτά μπορούν να στηρίξουν το ένα το άλλο. Εδώ λοιπόν θα ε, αναφερθώ στις βασικές αρχές του ε, Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και θα ήθελα να εξετάσω και πώς εφαρμόζεται, πώς έχει γίνει αποδεκτό από τα κράτη-μέλη και τέλος θα αναφερθώ σε κάποια ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση του πλαισίου με την οδηγία. Καταρχήν όσον αφορά τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το πλαίσιο. το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων είναι ένα σημείο αναφοράς, ε, σαν ένας ε, πίνακας μετάφρασης, ένας τρόπος να συγκρίνει κανείς τα προσόντα, να γνωρίζει ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιο είναι το προφίλ των διαφόρων επαγγελματικών προσόντων. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι υπάρχει ε, αυξανόμενος αριθμός προσόντων στην Ευρώπη. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ποικιλομορφία και πώς μπορούν να συγκριθούν αυτά τα επαγγελματικά προσόντα μεταξύ του. Το πρόβλημα αυτό όλο ένα αυξάνεται. Προσπαθούμε λοιπόν να απλοποιήσουμε τον τρόπο που συγκρίνουμε τα προσόντα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ε, ε, διαμορφώνονται τα προσόντα στις διάφορες χώρες. Και δύο βασικοί στόχοι υπάρχουν ε, του ευρωπαϊκού πλαισίου. Ο ένας στόχος είναι να βελτιώσει την κινητικότητα, που είναι άλλωστε στόχος και της οδηγίας. Το άλλο είναι ο άλλος ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την κινητικότητα μεταξύ ε, τομέων. Για παράδειγμα, ε, και να, να επικεντρωθούμε στη διαβίω εκμάθηση. Ε, ε, διαβίω εκμάθηση πρέπει να, να συνδυάσει κανείς, για παράδειγμα, την πρακτική εμπειρία με την επίσημη μάθηση. βασιζόμαστε σε 8 επίπεδα τα οποία βασίζονται στα λεγόμενα learning outcomes, τα αποτελέσματα της μάθησης. Και αναφερόμαστε στη γνώση, τις δεξιότητες ε, και την ε, ευθύνη, την ικανότητα. Το πλαίσιο καλύπτει το, όλο το φάσμα των ε, προσόντων από το Λύκειο μέχρι το υψηλότερο επίπεδο ακαδημαϊκής μόρφωσης. Έχουμε τους κύκλους που καθορίζει η διαδικασία της Μπολόνια. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε κατά νου τις αρχές της Μπολόνιας. Να μην καλύπτουμε όμως μόνο τις ακαδημαϊκές πτυχές, αλλά και την ε, πρακτική εμπειρία. Η αρχή των αποτελεσμάτων της μάθησης είναι πολύ σημαντική, διότι κατά παράδοση εκτιμούμε τα προσόντα ε, ανάλογα με ε, την ε, μάθηση, τη συνσφορά, δηλαδή το σε τι έχει εκτεθεί κανείς, αλλά εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα της μάθησης, δηλαδή τι, είναι, τι μπορεί να κάνει το πρόσωπο αυτό μετά το τέλος της εκπαίδευσης. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντική αλλαγή στον τρόπο που εξετάζουμε τα προσόντα. Τα 8 αυτά επίπεδα λοιπόν έχουν καθοριστεί με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πολύ δύσκολη δουλειά αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλουμε και σε εθνικό επίπεδο να ορίζουμε τις δεξιότητε ανάλογα με τα αποτελέσματα της μάθησης. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τη διαφάνεια, αυτό έχει σοβαρή συνέπειες όσον αφορά τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα. Ποιες λοιπόν είναι οι βασικές ημερομηνίες και προθεσμίες. Η σύσταση για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ε, υπεγράφει στις 22 Απριλίου του 2008 και έχουμε δύο βασικές προθεσμίες. Το 2010 οι χώρες ε, καλούνται να ε, αναφέρουν ε, τα εθνικά επίπεδα ε, δεξιοτήτων στο EQF και το 2010 θα πρέπει να έχουν αναφέρει σχετικά με τα πιστοποιητικά και διπλώματά τους. Παρακαλώ, αλλάξτε διαφάνεια, λέει ο μιλητής. Ποια είναι λοιπόν η παρούσα κατάσταση και είναι σημαντικό αυτό διότι δείχνει πώς γίνεται αποδεκτό αυτό. Πώς βλέπουν τα, κράτα, τα κράτη-μέλη τη χρησιμότητα του EQF. Τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων που αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά την κατάσταση του ευρωπαϊκού πλαισίου. 27 κράτη-μέλη ε, ε, ε, έχουν πει ότι θα έχουν ε, υποβάλει τι αναφορέ του στο EQF μέχρι το τέλο του 2011. Αυτό είναι μια χρονιά καθυστέρηση σχέσης σε σχέση μέχρι το 2010. Παρ' όλα αυτά είναι θετικό. Και κοιτάμε και άλλε χώρε όπω είναι η Αυστραλία και ο Καναδά και νομίζω ότι βλέπουν ότι είναι πολύ λογικός τρόπο να συγκρίνει κανεί προσόντα αυτό. Το EQF είναι ε, προαιρετική διαδικασία, αλλά ε, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς ε, κρατών μελών και επίσης και από τρίτες χώρες. Τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και την Οδηγία 2005-36. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα δούμε ως συμπληρωματικά μέσα. Αν επικεντρωθούμε στην ε, διαφάνεια και την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε. Πρόκειται για μια ενίσχυση ε, της βάσης. Σημαντικό είναι να προσέξουμε ότι το ΙΚΙΟ κάνει κάτι παραπάνω. Επικεντρώνεται στην μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, επικεντρωνόμενο στην διαφάνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό σε μια προαιρετική διαδικασία, μια θεωρητική διαδικασία κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να πούμε, και αυτό αναφέρεται πολύ σαφώς στην σύσταση του EQF, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2008, Σημαντική είναι λοιπόν η νομική βάση. Ο ρόλος του EQF είναι να βελτιώσει την ποιότητα, την εμπιστοσύνη και να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας. Με την επικέντρωση στα αποτελέσματα της μάθησης, έχουμε ένα στοιχείο πολύ χρήσιμο για την, ε, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Eh Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες ε, ε, οι οποίοι μας παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία και που κράτησαν και το χρόνο. Σας ευχαριστώ γιατί μας παίζει ο χρόνος. Θα σας πρότεινα τώρα να δείσουμε μεταξύ μας για 25 λεπτά. Υπάρχουν ε, έξι άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε τις παρεμβάσεις ε, με μιας και στη συνέχεια να απαντήσουν οι προγνώσεις και θα δώσουμε και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επικεφαλής της ε, αρμόδιας μονάδας της ΓΑΜΑ αγοράς. Κύριο Σουάπ, θέλετε να κάποιο σχόλιο να σας ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την Προεδρία σας κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης. Ευχαριστώ πολύ και όλους όσους πήραν τα λόγο, γιατί μας δίνουν ένα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, πλαίσιο για τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το θέμα των επαγγελματικών προσόντων. Η εσωτερική αγορά σαφώς και λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν είναι πάντα ομαλός το θέμα αυτό. Και βεβαίως θα προσπαθήσω εδώ να μιλήσω για ένα από τα επαγγέλματα. Μιλήσατε κι εσείς για τους νομικούς, για τους ε, δικηγόρους και σαφώς και πάντα το θέμα αυτό είναι δύσκολο να το δούμε συλλογικά. Εσείς κάθε φορά που αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα το βλέπετε ατομικά υπάρχουν περιπτώσει που μπορεί να καλύπτουν πολλέ. ε, Καλύτερα να ακουστούν όλες οι ερωτήσεις. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στον κύριο Μπιόνεβολτ θα ήθελα να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παρουσιάσετε τα πράγματα και εμείς νομίζω στο άρθρο 11 συζητήσαμε στο άρθρο 11 της οδηγίας για την αναγνώριση των προσόντων το θέμα δηλαδή της διαβίου κατάρτισης, της επαγγελματικής κατάρτισης. Μήπως θα ήταν δηλαδή διαφορετικός ο τρόπος ταξινόμησης Ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχει το σύστημα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ κάνω μία ερώτηση, αλλά ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να το απαντήσει. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια έκθεση του 2012 και βεβαίως περιμένουμε εξελίξεις στον τομέα αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που θέσατε. Στην αρχή ακούγοντάς σας, χάρηκα θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν δυσκολίες και όλα πάνε καλά. Βεβαίω, όταν μπαίνει κανεί σε πιο ειδικέ περιπτώσεις συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν ε, δυσκολίες όσον αφορά τους μηχανικούς παραδείγματο χάρη. Το θέμα τη πλατφόρμας ήταν μια ιδέα που αρχικά είχε θεσπιστεί για τους μηχανικούς. Τελικά βλέπουμε όμως ότι δεν προχώρησε. Η επαγγελματική κάρτα ενδεχομένως θα ήταν μία λύση. Αλλά και αυτό θα πρέπει να το επανεξετάσουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι το μέλλον θα εξαρτηθεί από τέτοιου είδους ιδέες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ακούσω όλους όσους μας κάνατε παρουσιάσει για το θέμα αυτό, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μία απάντηση. Κύριε Μέτσλερ, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Όπως και ο Ανδρέας Φάπ. Κάθε φορά μιλάμε για ειδικέ περιπτώσεις που δημιουργούν πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, η άδεια για την εγκατάσταση ενός κομωτή. Ξέρετε ότι στη Γερμανία υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη, αν θέλετε, ρύθμιση αυτού του επαγγέλματος όσον αφορά την εγκατάσταση και την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν εάν υπάρχουν ρυθμίσεις συλλογικέ ή αν κάθε φορά προκύπτουν σε ατομικό επίπεδο τα προβλήματα αυτά και λύνονται σε ατομικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάιλερ. Κάθομαι σε λάθος θέση, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να πάρω το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι πολλές ενώσεις με τις οποίες μίλησα έχουν πει το εξής. η σημερινή συζήτηση δεν είναι ε, βήμα για την αναθεώρηση της ε, οδηγίας. Ε, δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα γίνει αναθεώρηση. Αυτό μπορεί να το συζητήσουμε σε 3 τεσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. Αλλά πάντως δεν είναι προγραμματισμένο, αυτό θα το δούμε μαζί με την Κομισιόν. Πριν λίγες εβδομάδες λάβαμε την ανάλυση που έχει να κάνει με το πού βρίσκονται τα προβλήματα τα κράτη-μέλη έχουν ακόμα μεγάλη καχυποψία το ένα απέναντι στο άλλο. Ο καθένα θεωρεί ότι έχει το καλύτερο σύστημα, όλοι οι άλλοι χειρότεροι και δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν να μπει στα χωράφια μα. Ο Γερμανό ε, ομιλητή ε, πολύ ωραία μίλησε για ένα μέτρο ε, εκφοβισμού. Να υπάρχει δηλαδή ένα είδος ένα είδο προστατευτισμού, να θέτουμε τον πύχη τόσο ψηλά ώστε να μην μπορεί να το φτάσει κανείς άλλος. Εγώ Αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει προχωρήσει περισσότερα το θέμα των ε, πιστοποιητικών ε, που ε, θέλει να εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί σας. Και η βιομηχανία τι κάνει σχετικά. Ε, θεωρώ ότι δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα ακόμα. Επίσης, ε, όσον αφορά τους γιατρούς, υπόθηκε ότι θα είναι χρήσιμο να υπάρχει μητρό παραβάσεων, ώστε οι ασθενείς ε, να μπορούν ε, να λαμβάνουν σχετικέ πληροφορίες. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο για τους αρχιτέκτονες, για παράδειγμα, όταν θέλει να χτίσει κανεί ένα σπίτι. Ε, όταν όμως μιλάμε για γιατρούς, το κράτος έχει την αρμοδιότητα σχετικά με την πιστοποίηση των γιατρών και αν κάποιος έχει ένα τύχημα, αν κάποιος αρρωστήσει, δεν μπορεί πρώτα να, κάτσει, να δει αν είναι, ε, αν είναι ο γιατρός του. Και μία τελευταία παρατήρηση. Δεν θέλω να μιλήσω για τους ε, ξεναγούς. Και εγώ ξέρω αρκετές ε, τέτοιες περιπτώσεις. Αρκετοί έχουν στραφεί προς μένα. Ιδιαίτερα όσοι πήγαν στην Ιταλία και δεν μπορούσαν να εργαστούν εκεί, ενώ δεν το ξέρανε από πριν. Η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με τη συνεργασία. Σημαντικό θέμα όχι μόνο σε σχέση με την οδηγία για τις ε, υπηρεσίες, αλλά και με τούτη, ε, σε σχέση με τούτη την ε, οδηγία. Σημαντικό είναι να υπάρχει μια πλατφόρμα ώστε να γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Δεν θέλουμε να ξαναγκάσουμε τα κράτη-μέλη, δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν ε, την ε, να εναρμονίσουν τα πάντα και ε, ας το κάνουν αυτό τα κράτη-μέλη. Να μην έρθει κανεί να πει ότι το κοινοβούλιο το έκανε. Μια πλατφόρμα βέλτιστων πρακτικών λοιπόν θα ήταν πολύ χρήσιμη. Γιατί δεν λειτουργεί αυτό κατά τη γνώμη σα. Ε, Μήπω μπορεί να απαντήσει και η Κομισιόν σε αυτό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Ε, πραγματικά ήταν πολύ ενημερωτικό αυτό το απόγευμα. Εύχομαι ήταν εδώ περισσότεροι συνάδελφοι να σα ακούσουν. Ο κ. Μέτσλερ ε, αναφέρθηκε ε, στη Solvit και θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο για ποιες είναι οι εμπειρίες των υπολείπων με το Solvit ο κύριος Φιλίπ ε, τώρα από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο αναφέρθηκε σε ένα ποσοστό των γιατρών και είπε ότι ε, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλήσατε για ανισορροπία, για την ασφάλεια των ασθενών και για το, ε, την πρόσβαση στο επάγγελμα. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα στο εκατό ε, για μια χώρα που σας δίνει επαρκείς πληροφορίες, παραδείγματος χάρη για ένα συγκεκριμένο άτομο. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν παραδείγματος το θα εγκρίνεται ένα γιατρό από μια άλλη χώρα, τότε εσείς έχετε το άχθος τελικά που θα τον ε, εγγράψετε, γιατί εσείς τελικά είστε η αρμόδια ιατρική αρχή και αν τελικά προκύψει ότι το άτομο αυτό έχει κάνει λάθη σε άλλες χώρες, ε, τελικά πώς παρεμβαίνει η GMC. Εσείς θέλετε να υπάρχουν όλες οι πληροφορίες διαθέσιμες για να μπορείτε να λάβετε μια σωστή απόφαση. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και στα 27 κρατημέλη, αν κάποιος παίρνει το χάρη, γιατρός ή σε κάποιο άλλο επάγγελμα δεν ε, είναι ικανός και δεν θα πρέπει να ασκεί το επάγγελμά του. Και αυτό, αναφέρω, αυτό, σε αυτό αναφέρουμε σε ένα γιατρό είτε από το Ηνωμένο Βασίλειο είτε από άλλες χώρες και θα ήθελα να θέσω και μια ακόμη ερώτηση. Όταν ε, αναφέρεστε στο άρθρο 53, ε, το άρθρο 53 αναφέρεται στη γνώση των γλωσσών και αναρωτιέμαι πόσοι γιατροί συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εράσμους. Επίσης, ε, για τον ε, κύριο Τζένσερσον και για τις ε, διάφορα προσόντα. Και εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα με τη Γερμανία. Παρ' χάρη, δεν υπάρχει επαρκή αναγνώριση των προσόντων. Ε, κάποιοι άνθρωποι μεταβαίνουν στη Γερμανία και δεν μπορούν να εργαστούν εκεί. Γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ. και ελπίζω εδώ ε, κανείς ε, τελικά να μην ασκεί με λάθος τρόπο το επαγγελμά του. Πάντως σας ευχαριστώ και αναμένω να ακούσω τις απαντήσεις σας. Merci. Ευχαριστώ. Κύριος Άμπορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Χάρμπορ. Να σας ευχαριστούμε και για αυτή την ε, πολύ καλή ακρόαση. Θα ήθελα να φερθώ σε κάποια θέματα και ίσως ε, να εκμεταλλευτούμε το ότι έχουμε τους εμπειρογνώμονες εδώ για να μας δώσουν κάποια καθοδήγηση για το οποίο πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες ε, της Επιτροπής μας. Καταρχήν, να πω ότι εμείς ε, ως ε, άτομα που γνωρίζαμε ήδη έχουμε παραγγείλει μια μελέτη για το θέμα αυτό και αρκετοί που σας την καλωσορίζετε και εκεί αναφερόμαστε σε αρκετά θέματα που φορούσαν την εφαρμογή της εφιστάμενης οδηγίας. Κάποιοι είπαν ότι το βασικό πλαίσιο της είναι εύρωστο, αλλά τα εργαλεία εφαρμογή ίσω δεν έχουν απτυχθεί τόσο καλό όσο θα έπρεπε. Και υπάρχει γι' αυτό το σημαντικό θέμα των σχέσεων και τη ανταλλαγή πληροφοριών. Εκεί θέλετε να υπάρξει βελτίωση. Και νομίζω ότι αυτό φυσικά πρέπει να το κάνουν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν πρέπει να τα βοηθήσει, γιατί μιλάμε για ένα σημαντικό τομέα της μεταφοράς της νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο. Όμως ε, είναι καλό να υπάρχουν κάποιες συστάσεις σε αυτόν τον τομέα και θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το αν συμφωνείτε με τα συμπεράσματα της μελέτης μας ε, και πώς μπορούν ε, να υλοποιηθούν. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα της εμπιστοσύνης προέκυψε πολλές φορές για το πώς δηλαδή μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη Εδώ έχουμε κατά νου τη δυνατότητα η Επιτροπή μα να καλέσει μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου να έρθουν και να μα αναφέρουν τι δικέ του εμπειρίε, γιατί θεωρούμε ότι ε, αυτό το θέμα ενδιαφέρει και ε, του εθνικού βουλευτέ, γιατί νομίζω ότι έχουν εμπειρίε, επειδή μπορεί να είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο, αυτό σχετίζεται κυρίω σε σχέση με ο κ. Δεμπρούστα, για την αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματικών προσώπων προϊόντων και την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Και φυσικά αυτό συμπίπτει και με τη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο τη οδηγία των υπηρεσιών, που είναι τον επόμενο μήνα. Και ένα από τα θέματα που έχουμε στην οδηγία των υπηρεσιών είναι το θέμα των ε, προτύπων ποιότητα στι διασυνολογικέ υπηρεσίε. Ε, εγώ νομίζω ότι ο τουρισμό ήταν ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για τι διαφορέ που βλέπουμε στι εθνικέ προσεγγίσει. Δηλαδή, σε ορισμένε χώρε ε, οι πράκτορε πρέπει να έχουν εγγραφεί σε εθνικό επίπεδο, σε άλλε χώρε όχι για να παράσχουν αυτέ τι υπηρεσίε. Εγώ νομίζω ότι κατά την αθεώρηση τη νομοθεσία, αμφισβήτητα θα προκύψουν να αυτά τα προβλήματα. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέτε εσείς για το τι μπορεί να γίνει. Γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σαφής ευκαιρία για τα επαγγέλματα που αναγνωρίζονται ε, όμως ε, σε ορισμένες χώρες αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε πρακτική απέτηση και ίσω αυτό θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με κάποιο διασυνοριακό πρότυπο, το οποίο θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν οι καταναλωτέ. Αν πούμε δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ότι ακόμη και σε μια χώρα που δεν υπάρχει νομική απέτηση, απαιτούμε, παραδείγματο χάρη, να υπάρχουν κάποια πρότυπα για του ταξιδιωτικού πράκτορε, αυτό θα ήταν καλό και για του επαγγελματίε, αλλά και για του καταναλωτέ. Και πρέπει να δούμε πώ αυτό σχετίζεται με το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Και γύρω στο 2011 θα τα δούμε δούμε όλα αυτά εννοείται όταν θα έχουμε ε, υλοποιήσει την εξέταση νομοθεσία, θα έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και θα έχουμε και μια εικόνα πλήρη τη οδηγία. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σύνολο παραγόντων που θα εμφανιστούν από κοινού. Και τελική ερώτηση πώς ε, δημιουργούμε ε, μια συντονισμένη και λογική απάντηση σε όλα αυτά που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί ε, νιώθουν ότι έχουν δικαίωμα να μπορούν να εργαστούν και να μετακινηθούν και να ζήσουν σε άλλες χώρες και τελικά πώς βοηθούμε τους καταναλωτές. Πρέπει να τους δώσουμε σαφείς ενδείξεις ε, για την ε, ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρουν τα άτομα αυτά και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως στον τομέα της υγείας. Και ε, πώς ε, θα ενθαρρύνουμε ε, το όλο πλαίσιο όταν έχουμε το σχάρι κάποια μέσα τα οποία είναι κούσια και άλλα που είναι υποχρεωτικά. Νομίζω ότι ε, η Επιτροπή ήθελε να ξεκινήσει από νωρί ε, τη συζήτηση και στη συνέχεια να δούμε αν μπορεί να υπάρξουν ε, ορισμένα συγκεκριμένα θέματα που θα θέλουμε να προωθήσουμε του επόμενου 18 μήνε μέχρι την αναθεώρηση που θα κάνει η Κομισιόν, που ίσω θα μα αναφέρει σε λίγο. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όλοι έκαναν ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα τους. Καλό θα ήταν λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά να πάρετε το λόγο και σε ένα 1,5 λεπτό να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας αφορούσαν. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω στην κυρία Γκέπχαρτ καταρχήν. Αυτό που συμβαίνει από το 2005 μέχρι σήμερα, τα κράτη-μέλη όντως προόδευσαν στο θέμα της περιγραφής και του ορισμού αυτών των προσόντων και υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μία εξέλιξη σήμερα σαφώς και έχει αλλάξει ακόμα και η νοοτροπία που αφορά το θέμα αυτό. Και αυτό είναι κάτι που σαφώς και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω σύντομα στον κύριο Χάρμπορ, ο οποίος αναφέρθηκε στον δικό μας τομέα. Είπα στην παρουσίασή μου ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες σαφώς και επηρέασε περισσότερο τον κλάδο μας από ότι η οδηγία για τα προσόντα. Παραδείγματος χάρη, μετά την μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η Γαλλία απλοποίησε την νομοθεσία για τους ε, ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους tour operators. Ξέρετε, η Γαλλία είναι πολύ καλή όσον αφορά το περίπλοκο νομοθετικό οικοδόμημα. Το κατάφεραν λοιπόν. Η Ισπανία επίσης αλλάζει την νομοθεσία της. Η Ελλάδα εξετάζει την νομοθεσία της για το θέμα αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας μεγάλος αριθμός κρατών μελών σταδιακά συγκλίνουν σε κάτι που ενδεχομένως κάποια μέρα θα γίνει η κοινή πλατφόρμα όσον αφορά την πρόσβαση και τις κοινέ δεξιότητες και προσόντα των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Υπάρχει από τη μία το πακέτο, το οποίο ενδεχομένω θα αναθεωρηθεί του χρόνου, ακούμε, έτσι μας λένε από την Επιτροπή, και το πακέτο το οποίο επιβάλλει μία σειρά υποχρεώσεων ε, στους ταξιδιωτικούς πράκτερους όταν πολλούν τουριστικά πακέτα, ταξιδιωτικά πακέτα στους πελάτες τους. Την ίδια ώρα ξέρουμε ότι τα δικαιώματα, η προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών είναι υπό αναθεώρηση, κάτι που θα επηρεάσει επίσης το δικό μας τομέα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι κάποιοι από τους βουλευτές που πήραν το λόγο μίλησαν για αυτή την επαγγελματική κάρτα. Σαφώς και είμαστε υπέρ για τους ξεναγούς, είμαστε σαφώς υπέρ και για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, για τους tour operators, όπως είπα και αρχικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επιληθούν διάφορα προβλήματα που μας αφορούν σήμερα. Merci ευχαριστώ θα απαντήσω σε δύο σημεία. Καταρχήν το Solvit και την ερώτηση της κυρίας Γκέπχαρτ. Γιατί η κοινή πλατφόρμα δεν προχώρησε. Εμείς αρχικά βασιστήκαμε σε μια ιδέα που ήταν και η ιδέα της Επιτροπής ότι υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα για τους μηχανικούς. Ένα επάγγελμα δηλαδή. Τελικά όμως είδαμε ότι όταν μπήκε αυτή η ιδέα στην κοινή πλατφόρμα με την οδηγία, τα κράτη, οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών θα έπρεπε να δεχτούν ήδη όλους τους μηχανικούς που ανταπακρίνονταν στα κριτήρια αυτής της κοινή πλατφόρμας. Ένας χημικός μηχανικός όμως μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του στα πλαίσια αυτής της κοινή πλατφόρμας στον τομέα ενός πολιτικού μηχανικού. Σαφώς δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια ρύθμιση. Αυτό που θέλαμε είναι να αναγνωριστούν τα προσόντα ενός συγκεκριμένου ατόμου σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτό λοιπόν που είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η οδηγία είναι ότι φόβησε τα κράτη-μέλη και στη δεύτερη ανάγνωση, στο άρθρο 15, υπήρξε μια διαφοροποίηση που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα για το κάθε επάγγελμα. Για τους χημικούς μηχανικούς μία πλατφόρμα, για τους πολιτικούς μηχανικούς μία άλλη κτλ. Και ήδη υπάρχουν 20 σήμερα τέτοιες ε, δυνατότητες δημιουργίας μιας κοινή πλατφόρμας. Άρα το πέρασμα από τον ένα τομέα στον άλλο δεν μπορούσε παρά μόνο να γίνει με την κοινή πλατφόρμα. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που δεν προχώρησε. Σιγά σιγά θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια ιδέα και δεν μπορούμε που δεν λόγο να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη μια τέτοια επαγγελματική κάρτα. Αυτό μπορεί να κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που εγγράφονται σε αυτή την επαγγελματική κάρτα λαμβάνονται υπόψη από το κράτος μέλος, τη ρυθμιστική αρχή και να μην απαιτούνται επιπλέον στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά. Τώρα, όσον αφορά το Solvit, εμείς την Ομοσπονδία λαμβάνουμε κάθε είδους προσφυγές, διαμαρτυρίες για μηχανικούς παραδείγματος χάρη που θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα και είναι, έχουν σπουδάσει στην Αγγλία. Κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν αναγνωρίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα το Βρετανικό στην Ελλάδα. Προσπαθούμε λοιπόν να ρυθμίσουμε μέσω του Solvit, δεν είμαστε όμως σε επαφή άμεση με τα άτομα και ε, η επαφή μας γίνεται μέσω των επαγγελματικών ενώσεων και συλλόγων. Δεν έχουμε λοιπόν όλες τις πληροφορίες. Ο κύριος Μέτσαρ. Κυρία Πρόεδρε, ε, καταρχήν να απαντήσω στον κύριο Σβάπ. δεν είναι σύμπτωση το ότι θέλετε να δημιουργήσουμε ομάδες, ούτε ε, θα ήθελα να ε, σας ε, κατηγορήσω ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι λάθος, αλλά φυσικά θα πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση. Κυρία Κέπχαρτ. Εσείς ρωτήσατε για τους κομμωτές. Ε, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ελπίζουμε και το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων ε, επαγγελματικών προσόντων είναι ε, πολύ σημαντικό μέσο για αυτό. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά για να πείσουμε τον κόσμο ώστε να έχουμε και αποτελέσματα από την εκπαίδευση. Δυστυχώς θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σχετικά με την ποιότητα των εξετάσεων, διότι η πείρα μου μου δείχνει στη Γερμανία και μόνο ότι ανάμεσα στα διαφορετικά κρατήδια γίνονται συνέχεια πολλές συζητήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, εξετάσεις στο τέλος του Λυκείου. Θα ήταν καλό να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι έτσι ίσως να έχουμε μια πιο γρήγορη ε, απάντηση. Κυρία Βάιλερ, μιλήσατε για την ποιότητα. Αυτό είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η καχυποψία των κρατών μελών μεταξύ τους και αυτή η καχυποψία περνάει και στους πολίτες. Κανένας ε, δεν αμφισβητεί την ποιότητα της δική του δουλειά. έχει όμως καχυποψία απέναντι στους άλλους. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει διαφάνεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους πόρους, περισσότερο δυναμικό στην επικοινωνία. Θα Πρέπει δηλαδή να εξηγήσουμε γιατί ε, κάποιε εκπαιδεύσει διακούν περισσότερο λιγότερο κλπ. Με ρωτήσατε σχετικά με το Solvit. Με το Solvit έχουμε πολύ καλέ εμπειρίε. Ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να έχουμε ε, ενημέρωση σχετικά με το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Πολύ συχνά λοιπόν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα μέσω του Solvit. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κυρίως, Φιλίπ, νομίζω ότι σας έθεσαν και σας κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, Νομίζω ότι υπήρξε μια παρεξήγηση. Εμεί υποστηρίζουμε την αρχή τη κινητικότητας, τη ελευθερής κινητικότητας. Αυτό είναι σίγουρο. Όμω ε, όταν ε, ε, ουσιαστικά ε, κάποιος γιατρός ασκείται τα του μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που καταλήγουν και αυτό δεν μπορούμε να το αναγνωρίζουμε, να το παραγνωρίζουμε. Δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουν τα άλλα κράτη-μέλη με τις πληροφορίες που θα λάβουν για ένα γιατρό εμείς ε, ε, ουσιαστικά αυτές τις πληροφορίες τις δημοσιοποιούμε και στο κοινό. Μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση μέσω μιας ιστοσελίδας, όμως δυστυχώς δεν λαμβάνουμε τέτοια πληροφόρηση από άλλες ρυθμιστικές αρχές, κυρίως στην Ευρώπη. Και μπορώ να σας πω ότι περισσότερο έχουμε ε, με άλλες χώρες, οι Πολιτείε, Νέα Συλλανδία ε, και άλλες χώρες έχουν πολύ πιο διαφανή πολιτική από ό,τι παίρνουν το τόσο αλλα άλλα κράτη-μέλη. Οι σκανδιναβικέ χώρες είναι εξαιρετικέ ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών, ε, πάντοτε είναι διαφανεί και επιτρέπουν στου ασθενεί ή στου καταναλωτέ, αν θέλετε, σε αυτό το πλαίσιο να έχουν δυνατότητα να επιλέξουν ποιος θα είναι ο πάροχος ε, της πιο σημαντικής υπηρεσίας που θα λάβουν ε, ίσως ε, και είναι η ιατρική περίθαλψη. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να έχουν αυτό το δικαίωμα στην επιλογή. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει νομικό καθηκόν επί των νομοθετών και δεν θα πρέπει να υποσκάπτεται ε, ουσιαστικά από ε, τους επαγγελματίες και εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι οι γιατροί που έχουν ε, εγγραφεί ε, πρέπει να μπορούν ε, να θεωρούνται ότι προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σας πω ότι δεν ξέρω να σας απαντήσω για τον αριθμό των φοιτητών αλλά θα προσπαθήσω να μάθω τις και να επανέλθω. Μάλιστα, να κλείσουμε. Κυρία Λουσία Μέστρε, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, εμείς ε, εδώ είδαμε ότι υπάρχουν μία σειρά κολλημάτων και που δίνουν σε ρυθμισμένα επαγγέλματα, όμως τα προβλήματα υπάρχουν και μάλιστα πολύ σοβαρά προβλήματα έχουμε και σε επαγγέλματα που δεν ε, έχουν ρυθμιστεί, ούτε εντάσσονται στο πεδίο της οδηγίας και τα κράτη-μέλη τελικά μπλοκάρουν την είσοδο εργαζομένων ε, και τελικά αμφισβητούν ε, την εύρυθμη λειτουργία ε, της νέας αγοράς. Ε, αυτό είναι δραματικό και πραγματικά το έχουμε δει. Και έχει συμβεί και στην Πορτογαλία σε σχέση με ορισμένα επαγγέλματα. Εγώ νομίζω όμως ότι τώρα είναι κάπως πρόημο να αξιολογήσουμε το αντίκτυπο της οδηγίας 2036. Πράγματι, αυτή ήρθε για να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Ε, έτσι λοιπόν, ουσιαστικά ε, τελικά συγκεντρώνει αυτό ε, που είχαν προτιμήσει οι προηγούμενες επιτροπές σε επίπεδο γιατρών. Λουχαρίων τώρα θέλουμε να αποσαφηνίσουμε αυτά τα παραρτήματα, αυτή μπορεί να είναι ε, και η δουλειά των συντονιστών της ίδιας της Επιτροπής Αναγνώσης Επαγγελματικών Προσόντων. Αν λοιπόν κάτι τέτοιο, ίσως και όπως έγινε και για την ομάδα των αρχιτεκτών, δημιουργήθηκε μια συγκεκριμένη υπομάδα με πυρογνώμονα σε αυτό το τομέα για να δράσουν στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής. Έτσι λοιπόν, ε, εμείς ε, εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι συμβαίνει με την αυτόματη αναγνώριση ε, των επαγγελμάτων πρέπει στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή να εμπιστευτεί τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ε, που εντόπισαν ε, στα που έχουν ουσιαστικά αναφέρει στα παρτίματα ποια είναι τα απαιτούμενα για την αναγνώριση αυτών των επαγγελμάτων. Εγώ νομίζω ότι είναι ε, πολύ σημαντικό να εμπλέξουμε και το Solvit, αλλά να εμπλέξουμε και άλλα δίκτυα ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στο δίκτυο Cures, το οποίο μπορεί πράγματι να διασκεδάσει κάποιες ανησυχίες. Γιατί ο πολίτης όταν βλέπει, το χάρη, μία προσφορά θέσεις εργασίας χωρίς ε, στη συνέχεια να υπάρχει απέτηση αναγνώρισης, ε, μπορεί τελικά να χάσει κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμά του. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη διάδοση των πληροφοριών και να συγκρίνουμε τα ωφέλη που έχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο με αυτά που αναγράφονται στην Οδηγία 2036. Σας ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης για την αγορά. Πιστεύω θα μπορέσετε κι εσείς ακούγοντας όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στα 10 λεπτά που σας δίνω να καλύψετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που δίνετε τη δυνατότητα να πω δύο λόγια. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που οργάνωσε αυτή την ακρόαση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις που ακούσαμε από τους ειδικού του τομέα. Θα ήθελα εγώ εισαγωγικά να αναφερθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι πολύ απλό. Σήμερα υπάρχει μία ε, οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε 15. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά περιορίστηκε σε μία. Μετά από πολλή συζήτηση. Αυτή η συζήτηση επιτέλους πιστεύω ότι τελείωσε. Η αναγνώριση των προσόντων των επαγγελματικών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που καλύπτει τρεις ελευθερίες. Ελευθερία εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών και ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Αναφερόμαστε πολύ συχνά σε μία από αυτές τις οδηγίες που ουσιαστικά δεν αναφέρεται στις τρεις ελευθερίες που σας προανέφερα, αλλά στις δύο. Μία οδηγία λοιπόν που καλύπτει προβλήματα, προβλήματα όμως που είναι πραγματικά προβλήματα που αφορούν ένα μικρό αριθμό ατόμων πλέον. Βεβαίως οι πολίτες, οι επαγγελματίες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες, για αυτούς το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Χάνουν τα πάντα, χάνουν την επαγγελματική τους ε, δραστηριότητα. Γι' αυτό λοιπόν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θεωρούν τα θέματα αυτά και τις δυσκολίες αυτές πάρα πολύ σημαντικές και είναι για αυτούς. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να οργανωθεί. Σήμερα δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα, βρισκόμαστε απλώς σε ένα από τα στάδια αυτού του οικοδομήματος. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα όπως αυτό της εσωτερικής αγαράς για την ανταλλαγή πληροφοριών, η ποσότητα αυξάνεται διαρκώς. 12.000 ε, τέτοιες ανταλλαγές πληροφοριών έχουμε σήμερα, κάτι το οποίο ήταν μόνο το 1 τρίτο στην αρχή της συζήτησης για αυτή την οδηγία πριν από τέσσερα χρόνια. Για ποια θέματα ανταλλάσσονται οι πληροφορίες, θέματα πειθαρχικών μέτρων, παραδείγματος χάρη, γιατί πολλές φορές ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να έχει αποτρεπτική ε, δράση, να λειτουργήσει σαν απειλή. Κάτι το οποίο βεβαίως μπορεί να απειλήσει προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων εδώ και των πληροφοριών. Δεύτερον, όσον αφορά αυτά τα πειθαρχικά μέτρα, οι αρμόδιες αρχές έχουν κάποιες δυνατότητες σήμερα και εδώ ε, στη συζήτηση που έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα ακούσαμε το θέμα της επαγγελματικής κάρτας. Πώς θα γίνει αυτό αποδεκτό στα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι υπάρχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από το ένα κράτος μέρος στο άλλο. Η ακροάση σήμερα δεν έδειξε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι υπέρ αυτής της επαγγελματικής κάρτας. Ξέρω ότι χρειάζεται λοιπόν πολύ σημαντική προσπάθεια ακόμα και πιστεύω ότι η εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό βήμα αυτό, αλλά έχουμε ακόμα πολλές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε καταρχήν ότι η απλοποίηση για όλες αυτές τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως έχει ξεκινήσει, θα υλοποιηθεί πραγματικά. Σήμερα αναφέρθηκαν δύο περιπτώσεις. Πρώτον, τα ιατρικά επαγγέλματα, η ασφάλεια των ασθενών. Τι γίνεται λοιπόν με την περίπτωση των ιατρών που ασκούν το επάγγελμα σε ένα άλλο κράτος μέλος. Βεβαίως χρειάζεται η ελευθερία άσκησης του επαγγέλματος για τους γιατρούς, αλλά χρειάζεται και η προηγούμενη, ε, αν θέλετε, ύπαρξη ενός πιστοποιητικού νόμιμης εγκατάστασης για τον κάθε γιατρό. Και αυτό είναι κάτι που σαφώς θα βοηθήσει στην διασφάλιση των ε, δικαιωμάτων του ασθενούς, της προστασίας του ασθενούς. 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ταξιδεύουν, είναι τουρίστες. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός και βλέπουμε ότι εδώ σαφώς και χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις για τον συνάδελφο που ανάφερε το θέμα αυτό. Πιστεύω το θέμα της προθεσμίας είναι κάτι που μας απασχολεί, αλλά σήμερα δεν είμαστε διατηθειμένοι να πάμε στην κατεύθυνση την οποία πρότεινε. οι τοπικές αρχές σαφώς εδώ θα πρέπει κάτι να κάνουν και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Το θέμα του κινητού στόχου, όπως αναφέρατε. Το θέμα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο τομέας αυτός εξελίσσεται διαρκώς. Μιλάμε για τα αποτελέσματα, μιλάμε για το περιεχόμενο αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θα πρέπει εδώ να δούμε τα κράτη-μέλη πότε θα μεταφέρουν αυτές τις διατάξεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η οδηγία για την αναγνώριση των ε, προσόντων συμπεριλαμβάνει και ένα πολύ παλιό ε, και εκτιμένο κάνοντας μια κατηγορία επαγγελμάτων για τα οποία αυτή η επαγγελματική κατάρτιση είναι προτεραιότητα. Εν πάση μιλήσατε για κινητό στόχο, συμφωνώ. Επίσης, μιλήσατε για αυτή την κοινή πλατφόρμα που απέτυχε, δεν λειτουργήσε. Να δούμε αν θα λειτουργήσει η επαγγελματική κάρτα. Αυτό εξαρτάται, επαναλαμβάνω, και από τις τοπικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει το εξή από εδώ και πέρα. Τέλος Νοεμβρίου θα δημοσιεύσουμε ένα εγχειρίδιο, έναν οδηγό, όσον αφορά τώρα την μεταφορά. Το επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση. Το 2011 είναι ένας φιλόδοξος στόχος. Επιτρέψτε μου να περιμένω τον διορισμό του Επιτρόπου για να σας πω αν το 2011 είναι η υλοποιήσιμο στόχος ναι ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι έχουμε μεταξύ ημών κάποια κοινά σημεία, σημεια κοινές διαπιστώσεις. Εδώ χρειάζεται εργασία, συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Συμφωνώ και με τον Μάλκομ, ο οποίος μίλησε για μια συνάντηση το 2010 με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ίσως αυτό να απλοποιήσει τα πράγματα, κύριε Ντεμπλουίστ. Ελπίζουμε η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας να αυξηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα Μιλήσατε για την έκθεση όσον αφορά την μεταφορά. Θα πρέπει βάσει του άρθρου 60 της οδηγίας να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Αν υπάρχουν βελτιώσεις, αυτό θα πρέπει να γίνει πριν το τέλος της εντολής μας και καλό θα ήταν να γίνει το 2013. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες, Ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι παρόντες. Υπάρχουν πολλοί που δεν είναι παρόντες, γιατί Δευτέρα πολλοί λείπουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.